Mes chers collègues, bonjour. Nous reprenons nos travaux, s'il vous plaît. Να ξαναξεκινήσουμε παρακαλώ στην άνθρωπο της εργασίας μας. Σήμερα το απόγευμα η Επιτροπή μας διοργανώνει μία ακρόαση δημόσια για τον αντικτύπο του Brexit στις ε, θαλάσσιες μεταφορές. Στόχος της ακρόασης αυτής είναι να ακούσουμε τους εκπροσώπους ε, του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, των μεταφορών, των λιμένων για το θέμα του Brexit, προκειμένου να καταλάβουμε στο βαθμό του δυνατού ποιοι είναι οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες των φορέων αυτών. Θα θέλαμε επίσης να ακούσουμε πώς οι εταιρείε του τομέα αυτού προετοιμάζονται για τον αντίκτυπο του Brexit και ποιες είναι οι ενδείξεις σε ό,τι αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου σε ό,τι αφορά τον τη μεταφορά επιβατών και προϊόντων, σε ό,τι αφορά μεταξύ την μεταφορά μεταξύ της Υπηρετικής Ευρώπης, της Ιρλανδίας και, του Ηνωμένου, και της Αγγλίας. Θέλαμε να ακούσουμε λοιπόν την απόψη των διαφόρων αυτών φορέων του κλάδου και τι θα θέλαμε να περάσουν ως μήνυμα προς τους διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ακρόαση θα λάβει χώρα σε δύο μεγάλα τμήματα. Στο πρώτο τμήμα θα ακούσουμε τους εκπροσώπους των μεταφορέων. Στο δεύτερο μέρος θα συζητήσουμε με τους εκπροσώπους των λιμένων. Και κάθε πάνελ θα ακολουθείτε από γύρω ερωταπαντήσεων. Καλώς ορίσατε στους προσκεκλημένους μας, θα ήθελα να πω. Θα δώσω το λόγο λοιπόν καταρχάς ε, στους ε, ευρωβουλευτές που θα κάνουν μια εισαγωγή στο θέμα και να σας υπενθυμίσω ότι σε κάθε μέρος, ε, σε κάθε πάνελ, ο κάθε ο μιλητή θα έχει 7 χρόνια στην διάθεση του. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Μάρτιν Τόρσμαν, ο οποίο είναι γενικό γραμματέο τη ECSA, Ευρωπαϊκή, μάλλον Ένωση Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Πληκτητών. Να ευχαριστήσουμε επίση τον κύριο Μάρτιν Γκρίφιτ, ο οποίο είναι διευθυντή δημοσίων σχέσεων τη ε, Ένωση LIA για τη ακρογερόπλια και την κυρία Σου Μακένζη, διευθύντρια για την μετατροπή εταιριών και επιχειρήσεων από την P&O Ferries Ltd. Χωρίς να χάσουμε λοιπόν άλλο χρόνο, να δώσω το λόγο για 7 λεπτά στον κύριο Μάρτιν Ντόρσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και καταρχά να σας ευχαριστήσω που πήρατε την πρωτοβουλία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, όχι μόνο για τον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών, αλλά για όλη την οικονομία. Να υπενθυμίσουμε ότι δεν μιλάμε μόνο για τις θαλάσσιες μεταφορές και για τα λιμάνια. Μιλάμε για την όλη αλυσίδα από τους παραγωγούς, τους μεταποιητές, τους λιμένες, παρόχους υπηρεσιών, ε, καταναλωτές αν υπάρχει κάπου κάποια καθυστέρηση στις μεταφορές. Αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα. Καταρχάς, ό,τι αφορά την ΕΞΑ, την, ε, τον Ένωση Ενώσεων, αν θέλετε. Κοιτάξτε, κατάφερα να γυρίσω και τη διαφάνεια. Κάποιες ε, παρατηρήσεις ε, συναποτελούμαστε από 21 ενώσεις πλειοκτητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Νορβηγία Προσπαθούμε να προσπίσουμε τα συμφέροντά του και είμαστε στην... έχουμε δράση στις Βρυξέλλες, έχουμε νέα υπαλληλού. Δύο γενικές παρατηρήσει. Μία πρώτη παρατήρηση, κάτι που είπε ο κ. Κάσταλαΐν, ο οποίο είναι CEO του λιμένα του Ρότερνταμ. Πριν από δύο ημέρε δήλωσε το εξή. Οι κυβερνήσει προετοιμάζονται για το καλύτερο σενάριο, εμεί ε, προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο. Και αυτό θεωρώ ότι από την καλύτερη περιγραφή της κατάστασης για τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες για το ποια θα είναι η κατάσταση μετά την εμπορική συμφωνία, πώς θα τεμορφωθεί η πραγματικότητα. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε για το χειριστό σενάριο. Άρα έχουμε αφιερώσει πάρα πολύ ενέργεια και χρήματα στην προετοιμασία ενός σενάριου, γιατί δεν ξέρουμε τι είναι το χειριστό σενάριο στη τελική ανάλυση. Πολύ χρόνο έχουμε ταπανίσει. Άρα το βασικό ερώτημα που ρωτάμε και που θέλουμε να θέσουμε στις ομάδε ομάδες αμφότερες τη πλευράς να καταρτήσουν μια εμπορική συμφωνία, την καλύτερη δυνατή, αλλά το συντομότερο δυνατόν βασικά, για να είμαστε βέβαιοι για το τι θα μας φέρει στην τελική ανάλυση το αύριο. Έχουμε κάποιου μακροπρόθεσμους στόχους για να έχουμε ίσους όρους ανταγωνισμού εδώ στην Ευρώπη. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα φύγει από την Ευρώπη ίσως εμείς να έχουμε πιο πολλές ευκαιρίες να βελτιώσουμε το επιχειρηματικό κλίμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό από χώρες εκτός της Ένωσης. Αυτό θα αυξηθεί όταν θα φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο ενδεχομένω Άλλη μια ανησυχία, μάλλον κάτι θετικό. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι στην ίδια γραμμή όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο πολύ σε ό,τι αφορά τις Συμφωνία ελευθερίου εμπορίου για ανοιχτό και καθολικό εμπόριο και σε ό,τι αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο. Ενδεχομένω λοιπόν εδώ να έχουμε έναν σύμμαχο όταν μιλάμε για τον ΠΟΕ, τον ΩΣΑ, τον Διεθνή Οργάνωση Εργασία και τη Διεθνή Οργάνωση Εμπορίου. Τρει άμεσες προτεραιότητες. Καταρχάς σε ό,τι αφορά την ε, ελεύθερη μετακίνηση στην ε, θάλασσα και συνεχιζόμενη πρόσβαση στο τη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης ε, πρόσβαση στην ενέργεια. Να μην βρεθούμε σε μια κατάσταση που θα αποκλειστούμε από αυτά. Δεν λέω ότι θα συμβεί αυτό απαραίτητα, αλλά να το παρακολουθήσουμε. Κάποια αριθμητικά στοιχεία έχουμε στείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την παρουσίαση θεωρώ ότι είναι διαθέσιμη σε όλου, αλλά κοιτώντα τι εξαγωγές τη Ευρωπαϊκή Ένωση, 365 δι ευρώ από την άλλη πλευρά 170 δις ευρώ. Ένα εκατομμύριο, το ήταν το 93, τώρα είναι 4 εκατομμύρια φορτηγά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο βλέπετε ποια είναι τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ε, καθυστερήσεις για οποιοδήποτε λόγο, θα δείτε ότι είναι πραγματικά τεράστιες οι συνέπειες. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε τι σημαίνει αυτό. Έχουμε πλέον απόλυτη ελευθερία για τη μετακίνηση για τα φορτηγά από την Πρωτική Ευρώπη στην Ηνωμένο και και αντίστροφα. Και τα φέρει. Θα δείτε την κατάσταση μεταφέρει και λίγο αργότερα. Θα είναι διαφορετικά φυσικά τα πράγματα θα υπάρξει στην ελληνική διαδικασία εκ νέου. Στην Ολλανδία θα έχουμε πλέον 4,6 εκατομμύρια διαδικαστικές ε, δηλώσεις μάλλον τελωνιακές ε, κάθε χρόνο. Τα Ολλανδικά τελωνία σήμερα δηλώνουν ότι θα χρειαστούν χίλιες καινούργιους υπαλλήλου. Και οι κορυφαίες πέντε χώρες όταν μιλάμε για το εμπόριο μεταξύ ε, Ηνωμένου Βασιλείου και ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ολλανδία η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε την ελεύθερη μετακίνηση των, ε, του προσωπικού και των επιβατών. Αναγνωρίζονται φυσικά και από το Ηνωμένο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι σημαντικό να παραμείνει έτσι. Επίσης, σε ό,τι αφορά τους, το προσωπικό. Πολλές συμφέροντα που υπάρχουν ε, σε offshore ε, και το καθεξής. Είναι σημαντικό να μην αλλάξουν τα δικαιώματα τους για τους επιβάτες. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω τίποτα. Είναι πολύ οι άνθρωποι που μετακινούνται από και προ το Ηνωμένο Βασίλειο είναι εκτό Σέγγεν το Ηνωμένο Βασίλειο, ώρα έχουμε ήδη του ε, ελέγχου διαβατηρίων. Αν υπάρξουν όμω επιπλέον διαδικασίε, θα υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση. Τελευταίο. Διαφάνεια για τις περιορισμούς ε, στην πρόσβαση της αγοράς. Ως τώρα τα πράγματα είναι εντελώς ανοιχτά τα σκάφη μπορούν να ταξιδέψουν όπου θέλουν, εφόσον έχουν σημαία κράτους μέλους. Αν αλλάξει κάτι τέτοιο, ασφαλώς αυτό θα δώσει συγκριτικό πλεονέκτημα στα πλοία που θα πλέουν με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό προσφανώς δεν αποτελεί το σκοπό μας. Και στον τομέα offshore το ενωμένο Βασίλειο για το, για Βασίλειο η η Πρωτική Ευρώπη είναι σημαντική και εκεί απασχολούνται και πάρα πολλέ εταιρείε και σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρα, ε, παρουσίασή σας κύριε Ντόρσμαν. Με ουσιαστικά ερωτήματα είπατε πρέπει να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο. Ας προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε. Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Ο κύριος Γκρίφιτς έχει το λόγο για 7 λεπτά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας προσκαλέσατε να μιλήσουμε εδώ σήμερα. Η Ένωση Κροασγερόπλειων Είμαστε πολύ μικρό τμήμα ε, του, των θαλασσίων μεταφορών. Ε, αντιπροσωπεύουμε λιγότερο από το 1%. Ωστόσο, 5 εκατομμύρια ε, επιβάτες ε, μεταφέρουμε κάθε χρόνο και εκπροσωπούμε 150 ε, εταιρείε ε, που οργανώνουν κρουαζιέρες σε όλο τον κόσμο. Και άλλωστε και πολλοί ταξιδιωτικοί πράκτορες πολλούν εισιτήρια για κρουαζιέρες. Ε, όσον αφορά το σκληρό ή το πιο ήπιο ε, Brexit, είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς ε, τι συνέπειες θα έχει για τον τομέα μας. Ο τομέα των κρουαζιερών είναι ένα από του πιο κερδοφόρου όσον αφορά τι θαλάσσιες μεταφορέ. Το Brexit δεν θα έπρεπε να μα επηρεάσει πάρα πολύ δεν ε, θα αλλάξει τη δυνατότητα ε, των ε, πλοίων μας να ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για τα πλοία είναι ανοιχτέ οι θάλασσες και κινούμαστε σε ένα διεθνές νομικό πλαίσιο το οποίο δεν θα αλλάξει ακόμα και αν αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Brexit Επίσης δεν θα αλλάξει τη δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού στον τομέα μας. Δεν θα επηρεαστεί ε, η εθνικότητά τους ή ε, η διαμονή τους όταν βρίσκονται στο ε, σκάφος, στα σκάφη μας. Μπορεί να δυσκολευτούν κάπως περισσότερο οι βρετανικές επιχειρήσεις που απασχολούν Ευρωπαίους υπηκόου. Αυτή τη στιγμή έχουμε διάφορες γραμμέ που περνάνε και από το Ηνωμένο Βασίλειο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά με την αποχώρηση ε, του Ηνωμένου Βασιλείου ε, θα είναι σαν να επισκέφτονται το ε, Μαυροβούνιο ή την Ορβηγία ή την Τουρκία. Υπάρχουν κάποιες αβεβαιότητες τις οποίες θα πρέπει να μας βοηθήσετε να επιλύσουμε. Είμαστε προορισμός διακοπών και γι' αυτό ε, η μετανάστευση είναι μια από τις βασικές ανησυχίες μας διότι τι ε, περιορισμοί θα υπάρχουν για τις διάφορες πικότητες ε, όταν βγαίνουν στη στεριά. Και το ίδιο ισχύει για το προσωπικό μας. Οι θεωρήσεις τους και οι άδειες εργασίες τους πώς θα επηρεαστούν. Το η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν αρκετά σαφή. Ε, δεν θα αλλάξουν οι συνθήκες για κρουαζιερόπλια που επισκέφτονται το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά θα αλλάξουν οι τελωνιακέ ε, ρυθμίσεις ε, και πέρσι δημοσιεύτηκε λευκή βίβλος που δείχνει πώς μπορούν να επηρεαστούν. Ένα άλλο τομέα που μας αφορά είναι επιβάτες που αυτή τη στιγμή έχουν ε, ε, ενιαία προγράμματα ασφάλισης ε, ταξιδίου. Αυτό όμως θα αλλάξει αν αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη οι επιβάτες κλείνουν κρουαζιέρες για του χρόνου και θα πρέπει να γνωρίζουμε τι θα ισχύει για αυτούς που ταξιδεύουν και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουν να απολαύσουν όσο γίνεται καλύτερα τις διακοπές τους θα χρειαστούν θεώρηση για το ένα ή το άλλο μέρος. Ε, μάλλον όχι, αλλά χρειαζόμαστε βεβαιότητα ώστε να μπορούν οι ε, οι ταξιδιώτες ε, να λάβουν τα μέτρα τους. Επίσης, ε, θέλουμε να ξέρουμε κατά πόσο θα είναι καλοδεχούμενοι οι ε, τουρίστες ε, στι διάφορε χώρε Ο κύριο Φαρχόφστατ είπε ότι δεν θα έχουν αυτομάτως δικαίωμα να κάνουν τις διακοπές τους οι Βρετανοί στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είναι σωστό, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα ευγενικό. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να δούμε τι θα ισχύει για του επιβάτε μα. Πιστεύουμε ότι θα βολέψει και τις εταιρείες που οργανώνουν κρουαζιέρες και τους επιβάτες μας εάν ε, τα μέτρα που ισχύουν σήμερα συνεχίσουν να ισχύουν και για τους Βρετανούς μετά το Brexit, ε, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ασφαλίσεις. Επίσης, ε, ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να οργανώνουμε ε, ταξίδια με ενιαία ασφάλιση ταξιδιού. Προσβλέπουμε ε, στη συνέχιση των εργασιών πάνω στο θέμα αυτό τους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Γκρίφιθ για την παρέμβασή σας. Τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Μακένση. Έχετε το λόγο για 7 λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ονομάζομαι Σου Μακένζι, είμαι ε, υπεύθυνη των P&O Ferries και θέλω να, μάλλον ασχολούμαι με τα 11 λιμάνια από όπου λειτουργούμε και φυσικά με τη χρήση ε, υψηλής ε, τεχνολογίας. Προ-Brexit ήταν αυτός ο τίτλος. Εμείς ε, έχουμε 27.000 πλώες μεταξύ ε, Γαλλίας, Ιρλανδίας, ε, Αγγλίας, Ολλανδίας και Βελγίου. Και επίσης λειτουργούμε και με σιδηροδρομικά δίκτυα στην Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία και Ολλανδία. Δρούμε ε, και στην ε, Ρουμανία έτσι ώστε να προωθήσουμε τη μεταφορά των αγαθών από την Κίνα, από το δρόμο του μεταξιού. Πρόκειται για μια ιστορία 180 ετών όπου είχαμε μια δράση μεταξύ Νότιας Αγγλίας και η Βυρικής Χερσονήσου. Τώρα όμως ε, ασχολούμεθα με τις συνολικές ε, υποδομές εξαγωγών στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μιλάμε για φαρμακευτικά προϊόντα, ε, συγκεκριμένα προϊόντα, από λάδι, κρασί κλπ. κλπ. Έχουμε πολλούς εργαζομένους και είμαστε υπεύθυνοι για πλειάδα εργασιών που σχετίζονται με την επιμελητία και τους σιδηροδρόμους. Τη στιγμή που υπάρχουν αγαθά και επιβάτες μεταξύ Βρετανίας και Ευρώπης, θα έχουμε μία ε, υπηρεσία ποθμίων και επιμελητίας. Έχουμε ε, συνεργαστεί και με τις άλλες χώρες που συνεργαζόμαστε και με τους, ε, τομείς, τους διάφορους τομείς στο Ηνωμένο Βασίλειο έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις ε, του Brexit σε μας. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα περάσουμε στη συζήτηση για το πρώτο πάνελ εμπειρογνωμόνων Θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία ping-pong και μετά θα γίνει ένας δεύτερος γύρος όπου θα δώσουμε το λόγο στους συντονιστές πρώτα και μετά στο σύνολο των μελών. Πρώτος γύρος λοιπόν, αρχίζει ο πρώτος γύρος, για πέντε λεπτά θα έχει το λόγο ο καθένας ο κύριος Βίμ Βαντεκάμπ έχει το λόγο. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Και αντικαθιστώ σήμερα τον συνάδελφο Μάρκος Πίπερ, ο οποίος είναι ο ειδικό σε θέματα Brexit. Δυστυχώ έχει ανελημμένε υποχρεώσει. Και έτσι έχω και εγώ επιτέλου την ευκαιρία ω Ολλανδό θαλασσοπόρος που φοβάται το νερό να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση προς τον κύριο Ντόρσμαν. Είναι δύσκολη ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει επαρκώς τα προβλήματά σας και τα πρακτικά αυτά ζητήματα. Και να απαντήσετε το κατευθείαν. Παρακαλώ. Μάλιστα. Να απαντήσετε στα Ολλανδικά. στο Συμβούλιο ΑΞΑ είχαμε επίσκεψη εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εξηγήσαμε πώς έχει η κατάσταση και ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Προσπαθήσαμε να κάνουμε λοιπόν διάλογο. Έχουμε κάνει λοιπόν τρεις συνομιλίες ε, ως τώρα και ναι, έχετε την εντύπωση λέει κ. Φαντεκάμπο ότι τα καταλαβαίνουν. Κοιτάξτε, είναι διατεθειμένοι να ακούσουν. Ήταν πολύ διστακτική σε ό,τι αφορά την χορήγηση οποιασδήποτε ένδειξη... του πού θα κινηθούν τα πράγματα, αλλά μας εισακούν. Μία δεύτερη ερώτηση για τον κύριο Γκρίφιν και την κυρία Μακέντζη. Ο μοναδικός τρόπος για να σωθούμε είναι η μεταβατική περίοδος για να τα βγάλουμε πέρα. Δεν θα είμαστε έτοιμοι 31 Μαρτίου του 2019. Είναι ψευδέστηση αυτή. Κύριε Ντόρσμαν, Πώς αντιμετωπίζετε αυτή τη μεταβατική περίοδο. Είναι κάτι που σας απασχολεί, έχετε άποψη για το πόσο μεγάλα θα πρέπει να είναι, τι, τι, τι στοιχεία χρειάζεται. Κοιτάξτε, και αυτή η ερώτηση είναι πάρα πολύ δύσκολη για τη μεταβατική περίοδο. Θα πρέπει να ξέρουμε αυτή η μεταβατική περίοδο πού θα οδηγήσει, προ τα πού θα κινηθούμε. Θα είναι συνέχιση τη σημερινή κατάσταση. θα υπάρξουν αλλαγέ. Και αυτό έχει να κάνει και με την αβεβαιότητα που τόνισε αυτή εξ αρχή, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουν την κατάσταση οι επιχειρήσει. Γιατί πράγμα προετοιμαζόμαστε και η μεταβατική περίοδο. Πολύ σημαντική. Αλλά πώ θα με διαμορφωθεί και πόσο μεγάλη θα είναι, δύο χρόνια. από ό,τι μου φαίνεται αυτό είναι το μέγιστο όριο. Το, ε, δύο χρόνια θα είναι αρκετά σύντομη περίοδος, αλλά το βασικό είναι γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε, πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γκρίφιτ. Ε, συνομίλησα στο παρελθόν με την Τούι, που είναι συνάδελφος και ανταγωνιστής. Και όντω πρέπει να κλείσουν οι εισιτήρια για το 2019. Πώς θα το κάνετε λοιπόν αυτό, γιατί δεν έχουμε νομικό πλαίσιο στην παρούσα φάση. Όχι, συμφωνούμε μαζί ε, σα ότι ο κόσμο κάνει κρατήσει από πολύ νωρί για τα κρουαζιερόπλια, για τι κρουαζιέρε. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε και θα το παρακολουθούμε σε ό,τι αφορά και την μεταβατική περίοδο. Νομίζω ότι όταν οι επιβάτες μεταβαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ ευσυρε οι σχέσει λόγω έλευση Σέγγεν. Αυτό δεν θα αλλάξει. Θα αλλάξουν άλλα πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Ιδιαίτερα σε θέματα ασφάλεια ταξιδιού, ασφάλεια υγεία και το καθεξή. Ε, η κυρία Μακέντζη. Ναι, όντω μία μεταβατική περίοδο σίγουρα θα είναι ωφέλιμη και χρήσιμη. Συμφωνώ με του άλλου ομιλητέ για να καταλάβουμε προ τα πού κινούμαστε και γι' αυτό λοιπόν είναι δύσκολο να καθορίσουμε πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η μεταβατική περίοδο. Αλλά πιστεύω ότι η τεχνολογία αποτελεί το κλειδί για μια ομαλή μετέβαση. Όσο πιο σύντομα ξεκινήσουμε, τόσο καλύτερα. Χωρί μικρόφωνο, ο κύριο Να επανέλθω στον κύριο Ντόρσμαν. Ποια είναι η άποψη των Βρετανών στην ένωσή σας. Οι Βρετανοί στην παρούσα συμφωνούν στο ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν οι τρέχουσες ροές εμπορίου και παροχής υπηρεσιών. Το θέμα είναι τι θα γίνει και στο μέλλον σε ό,τι αφορά τι έδρε των εταιρείων κτλ. Αλλά σε ό,τι αφορά το εμπόριο, συμφωνούν απόλυτα και έχουν καλή επιρροή στη Βρετανική κυβέρνηση, ρωτάει ο κ. Φουμινκόμπ. Κοιτάξτε, να σα πω. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει στενή επαφή. Μάλλον ξέρω ότι υπάρχει στενή επαφή και αυτό είναι φετικό. Και οι εταιρείε φέρει συνομιλούν τακτικά με τι ε, Βρετανικέ αρχέ. Αυτή η ανταλλαγή λοιπόν απόψεων ε, πάει καλά. Το μεγάλο ερώτημα φυσικά είναι τι θα συμφωνηθεί τελικά. Το λέω και το ξαναλέω και θα συνεχίσω να το λέω. Τι συμφωνία θα επιτευχθεί από πλευρά Βρετανών. Θεωρώ ότι κάνουν ό,τι μπορούν για να βρουν στο συντομότερο δυνατόν τη σαφήνεια που χρειάζεται. Ο κύριος Γκρίφιτ μπορεί να απαντήσει στην ερώτηση για τους Βρετανούς. όχι, καλά. Εντάξει. Α, απαντάει. Ναι, συνεργαζόμαστε πολύ στενά με το επιμελητήριο το αντίστοιχο στην Βρετανία για να διασφαλίσουμε ότι όλα θα πάνε όσο πιο ομαλά γίνεται. Έχουμε καλέ σχέσει και με του εκπροσώπους των Βρετανικών Αρχών. να Ελπίζουμε έτσι να συνεχιστεί η πορεία αυτή. Μάλιστα. Και η κυρία Μακέντζε. Ναι, ακριβώ. Εργαζόμαστε πολύ στενά με τη Βρετανική κυβέρνηση και σε μεμονωμένο επίπεδο με το επιμελητήριο. Είναι πολύ επικοδομητική αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Η κυρία Άντερσον έχει το λόγο για πέντε λεπτά τώρα. Um, thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, μια γενική ερώτηση σχετικά με την, νομοθέτηση, την, την νομοθεσία, την νέα νομοθεσία και το γενικό πλαίσιο τους ε, κανόνες ε, ασφάλειας, για παράδειγμα, για τα επιβατικά πλοία. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Και όσον αφορά την αναγνώριση προσόντων επαγγελματικών προσόντων. Μια γενική ερώτηση προς όλους σας καταρχάς. Έχετε ανησυχίες σχετικά με το πώς αυτό θα λειτουργήσει ε, σε έναν κόσμο μετά το Brexit όσον αφορά την νομοθεσία. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν διεθνείς κανόνες, αλλά υπάρχει και συγκεκριμένη νομοθεσία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα πλαίσιο με το οποίο έχουν συμμορφωθεί όλοι. Τι ακριβώς θα γίνει στη συνέχεια. Ναι, σίγουρα. Είναι πολύ εύστοχο αυτό που λέτε. Αναφέρεστε στην ε, διεθνή νομοθεσία ε, όσον αφορά το περιβάλλον, για παράδειγμα. Εάν όμως χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να εισάγει επιπλέον νομοθεσία ευρωπαϊκή η οποία δεν θα ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε διότι αυτό σίγουρα μπορεί να επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα των ε, Ευρωπαίων εφοπλιστών. Αναφέρθηκα σε αυτό στην εισήγησή μου. Το νομοθετικό πλαίσιο σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε. Ναι, και νομίζω ότι όλα τα πλοία που ε, ε, λειτουργούν εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, που πλέον εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, πρέπει να συμμορφώνονται με του κανόνε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά βέβαια στο μέλλον, εάν δημιουργηθούν προβλήματα, θα πρέπει να το εξετάσουμε. Όπως ε, σας είπα ήδη, κινούμαστε εντό διαφόρων ε, κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να εφαρμόζουμε όλες τις ε, σχετικές οδηγίες. Η κυρία Άντερσον, σα ευχαριστώ πολύ. Δεύτερη ερώτηση όσον αφορά χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την καιροτομία, τι έρευνε ε, αλλά και τι υποδομέ. Έχετε εσεί ανησυχίε ότι μετά την αποχώρησή μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπάρξει απώλεια εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα αυτών και η ερώτησή μου απευθύνεται κυρίως στον κύριο Τόσμαν αλλά ίσως και στην κυρία Μακένζη. Μήπως μπορείτε να διευκρινίσετε λίγο. Η απώλεια χρηματοδότησης ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ήταν πολύ σημαντική για την ανάπτυξη νέων καυσίμων, πρόσβαση στην, ε, στις υποδομές, δημιουργία νέων υποδομών στο Ηνωμένο Βασίλειο το Ηνωμένο Βασίλειο ως προορισμός δεν θα είναι προβληματικό τώρα πια που θα είμαστε μόνοι μας όσον αφορά το επίπεδο επενδύσεων για παράδειγμα. Ναι. Αλλά εγώ σκεφτόμουν και όλας ότι θα υπάρχει κάποιο έλλειμμα με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Έτσι θα μειωθεί το ποσό που θα υπάρχει στη διάθεση κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα TNT. ο τομέας ε, των ε, θαλασσιών μεταφορών είναι διατεθειμένος για παράδειγμα να έχει πιο οικολογικό, πιο περιβαλλοντικά φιλικό στόλο και ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών αντιμετωπίζει δύσκολες οικονομικά εποχές. Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί λοιπόν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις και στην υποδομή. Η πρόκληση αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχει υγροποιημένο φυσικό αέριο σε όλα τα λιμάνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, και αυτό επηρεάζει τη δυνατότητα του να έχουμε πιο περιβαλλοντικά φιλικό στόλο. Ε, και μια τελευταία ερώτηση, κυρία Μακένζη. Ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε τον προηγούμενο μήνα ότι ε, οι Βρετανοί ναυτικοί δεν θα μπορούν να εργάζονται σε ευρωπαϊκά ε, σκάφη. Και φυσικά μας απασχολεί πολύ η προστασία των καλών προτύπων, ε, η διασφάλιση του προσωπικού και μάλιστα καλά εκπαιδευμένου φυσικού μπορεί να το, ε, ε, ε, εκπαιδευμένου προσωπικού μπορεί να το σχολιάσετε αυτό. ναι, το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να τα καθορίσουν αυτά και κατόπιν εμεί θα δούμε πώ θα εργαστούμε. Έχουμε προσωπικό όμω όλων των εθνικοτήτων ε, στα σκάφη μας. Δεν νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει σύντομα. Ε, η κυρία Άντερσον, δεν είμαι βέβαιη αν αυτό η αποτελεί απάντηση στην ερώτησή μου. Οι Βρετανοί ναυτικοί θα μπορούν να εργάζονται σε σκάφη με σημαία Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Μακένζη, φοβάμαι ότι δεν γνωρίζω την απάντηση αυτή. Δεν είναι αρμοδιότητά μου, αλλά μπορώ να το εξετάσω και να σα απαντήσω. Συνεχίζουμε με την κυρία Φώστερ. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι που δεν παρακολούθησα τον πρώτο παρουσιαστή, γιατί έχουμε παράλληλες ε, συναντήσεις. Ο Γκίφερ Χόφστατ δεν μιλάει για την ε, πλειοψηφία των μελών. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις και η Επιτροπή μας είναι πολύ παραγωγική. Έχω ασχοληθεί και συνεργαστεί με το Βρετανικό Επιτροπή επιμελητήριο με πολλούς συνεργάτες και είχα συναντηθεί με τους P&O Ferries για τον Μάρτιν και του Σου. Θα ήθελα να πω το εξής. Γίνεται μια δημόσια συζήτηση για να προωθηθεί το μέλλον αυτής της βιομηχανίας μετά το Brexit θέλουν να υποστηριχθεί η ανάπτυξη γιατί μιλάμε για 111.000 ε, θέσεις εργασίας και 50 δις στερλίνες για την οικονομία μας. Ε, ποια είναι η θέση σας ε, από τους δύο τομείς. Ό,τι περιορίζει τη, δυνατότητα δραστηριότητά μας προκαλεί προβλήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μετανάστευση. Θέλουμε να υπάρχουν ίσοι όροι δράσης παντού. Η χρήση της τεχνολογίας θα πρέπει να γίνεται για να μην υπάρχουν ε, έλεγχοι, περιττή έλεγχοι στα ε, λιμάνια. Αυτό και πρώτου Brexit, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία ακόμα περισσότερο για αγαθά που δεν προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να έχουμε απρόσκοπτες μεταφορές. Επόμενο σημείο και για τους δυο σας. Ορισμένοι ε, ε, εργαζόμενοι τομέα θεωρούν ότι ίσως θα πρέπει να γίνουν διμερείς συμφωνίες αυτό σε σχέση με τις ναυτιλιακές εταιρείες. Ως προς τη συνεργασία στην Ασία, για παράδειγμα, εγώ βρίσκομαι και στην αντιπροσωπεία Αυστραλίας, Νέας Ζηλανδίας και δεν έχουν κανένα πρόβλημα για διμερείς συμφωνίες για το εμπόριο. Θεωρείτε ότι θα έχουμε τις ε, δυνατότητες που θα ανακύψουν όταν εγκαταλείψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις P&O Ferries Σίγουρα υπάρχουν δραστηριότητες εντός ε, Ευρώπης, άρα δεν ασχολούμαστε με την Αυστραλία, με την Αυστραλία Νέα Ζηλανδία. Ναι, για τον ε, Μάρτιν. Για τον Μάρτιν είναι η ερώτηση. Παρόλο που θα ήθελα να... Παρόλο που θα ήθελα να πάω στην ε, Αυστραλία, ναι, όπως ξέρετε, τα κρουαζιερόπλια δρούν προς τα εκεί, γίνονται ταξίδια και θα εστιάσουμε την προσοχή μας και εκεί. Ναι, έγιναν ανακοινώσεις τύπου για τα κέρδη των συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου με άλλες χώρες για να αντισταθμίσει τις απώλειες δυνατοτήτων εμπορίου μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ήταν σαφές κατά πόσο θα υπάρξει αντιστάθμιση ζημιών. το τελικό αποτέλεσμα ίσως να είναι αρνητικό παρά τις διαπραγματεύσεις για συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Ευχαριστώ και για να απαντήσω γιατί έχω λίγα λεπτά. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη και δεν βλέπω μεγάλες αλλαγές μετά το Brexit. Θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις βεβαίως αλλά θα αντιπαρέλθουμε. Το ποτήρι είναι μισογεμάτο νομίζω και νομίζω ότι θα κρατήσουμε και πολύ καλές σχέσεις με τους φίλους και γείτονες. Σας ευχαριστώ πολύ που βρεθήκατε εδώ σήμερα από πλευρά της ομάδας CCR. Η κυρία Μάισνερ έχει το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε και να ευχαριστήσω όλους όσους μας μέλησαν εδώ. Θα συμφωνήσω με την Τζάκη Φώστερ, η οποία εκφράστηκε με μεγάλη αισιοδοξία και εγώ είμαι κανονικά πολύ αισιοδοξή και θα ήθελα πραγματικά να είναι το αποτέλεσμα αυτό που ελπίζουν πολύ αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν θα είναι έτσι. Είμαι από αυτούς που σκέφτονται όπως η Λουσί Άντερσον. Είπατε και ορισμένοι από εσάς αναφέρθηκαν σε καλές συνομιλίες με το Λονδίνο, με την Βρετανική κυβέρνηση, με θετικό κλίμα και είπατε ότι ήδη έχετε πει και στις Βρυξέλλες ε, τι θέλετε, αλλά δεν σας έχουν ακόμα υποσχεθεί τίποτα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και τα αρνητικά και να αναρωτηθούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες. Ε, προς την κυρία Μακέντζη συγκεκριμένα. Πολύ είναι η κυκλοφορία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρώπης ε, μέσα της μάχης. Υπάρχει η συνθήκη του 2013 για τις τελωνιακές διεκπαιρεώσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου και άκουσα ότι θα πρέπει να υπάρξει και ένας νέο, ένα νέο καθεστώς ε, μετανάστευση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε άποψη εσύ γι' αυτό. Απάντηση. Το άκουσα, προφανώς. Ε, και είναι θέμα της Βρετανικής και της Γαλλικής κυβέρνησης να βρουν τη λύση και προφανώ μετά να μειώσουμε τον αντικτύπο στι δράσει μα. Μάλιστα. Αυτό θα ήταν το πρώτο, αν αλλά θα μπορούσαν να παραμείνουν όσα έχουν, βέβαια. Για εσά θα ήταν καλό αυτό, αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν θα γίνει κάτι αυτό, γιατί υπάρχει ένα σύνορο στη μάχη. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια άλλη διευκρίνηση σε ό,τι αφορά τις ε, διατάξεις ε, δεν θα αλλάξει κάτι γιατί σε τελική ανάλυση υπάρχει ο διεθνής οργανισμός και αυτό ισχύει εξίσου και για τις δύο πλευρές αλλά θέλετε και είπατε ότι οι ναυτικοί θέλετε να έχουν ελεύθερη κυκλοφορία. Αυτό ασφαλώς και είναι το ευκταίο. Αλλά αν δεν ε, υπάρχει σήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Βρετανούς ε, ναυτικούς, τι θα σήμαινε αυτό για τις δικές σας ε, επιχειρήσεις. Και Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Για τις ε, συνθήκη τη διεθνή που υπάρχει για την εργασία και τις ε, διατάξεις της ε, Μπρίζ. Διεθνείς διατάξεις ισχύουν για όλο τον κόσμο είναι ένα διεθνές νομικό πλαίσιο. Αυτό δεν θα αλλάξει. Αυτό είναι σημαντικό. Σε ό,τι αφορά τώρα τις επαγγελματικές δεξιότητες. Σημαντικό θέμα αυτό. Αναγνωρίζουν τα κρατημέλη ε, τα διπλώματα και τα πτυχία των άλλων χωρών και τις επαγγελματικές ε, διατάξεις. Αυτό μας ανησυχεί. Θα πρέπει να συνεχιστεί. Οι Βρετανοί ναυτικοί που πλέον για παράδειγμα υπό Ολλανδική σημαία. Θα ήταν πολύ καλό να συνεχίσουν να μπορούν να, να ασκούν τις δραστηριότητες αυτές. Και αντίστροφα. Άρα ε, για τις διτάξεις της Μπρίζ έχουμε να πω ότι κατοχυρώνονται σε διεθνές πλαίσιο και βάσει αυτών η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναγνωρίζει τα διπλώματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί με το Ηνωμένο Βασίλειο αναγκαστικά. Ένα άλλο θέμα είναι κατά πόσον θα υπάρχουν ε, σχετικές, ε, αν υπάρχει σωστή ρυθμίση. Αν υπάρχει σωστή ρυθμίση δεν φοβάμαι καθόλου ότι θα υπάρξει θέμα. Δεν είναι προς το συμφέρον κανενός, καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλλη μια ερώτηση πάλι στον ε, κύριο Ντόσμαν, γιατί έχετε πολύ καλές ευχές. Μακάρι να εκπληρωθούν, είπατε, να υπάρχει ομαλή μεταφορά στη θάλασσα. Πού πιστεύετε ότι ενδεχομένως να υπάρχουν αυτές οι τριβές που φοβάστε. ενδεχομενω να στην παρατηρήση που έκανα για την αβεβαιότητα. Αβεβαιότητα. Για ε, το τι θα αλλάξει, αν θα αλλάξει κάτι, πότε θα αλλάξει, θα γίνουν έλεγχοι, θα καθιερωθούν έλεγχοι, σε ποιου τομείς ε, για θέματα υγείας, κτηνιατρικά. Έχουμε στην Ολλανδία 35.000 μόνο επιχειρήσεις ε, που θα πρέπει να καταβάλουν ε, δηλώσεις για το εμπορευμά του. Θα γίνουν αυτά ομαλά, πώς θα γίνει η μετάβαση, πόσο μάλλον αν υπάρχουν και επιπλέον προδιαγραφές. Όλα αυτά είναι ερωτηματικά. Τι θα μας φέρει το μέλλον. Merci beaucoup, Madame Meissner. Euh, Madame Vieux. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία... Yeah, ναι, όχι. Monsieur Kistelor, pour 5 minutes. Vous voulez pas... Ο κύριος Κίστελο για 5 λεπτά. Oh. Δεν θέλει να πάρει το λόγο. Ο κύριε Ροκέ. La parole est à vous pour 3 minutes. Oui, ah ben, j'ai pas... Δεν χρειάζομαι τρία λεπτά. Έχω μία απλή ερώτηση και προς τρεις παρεμβαίνοντας. Ποια ευεργετήματα προβλέπετε για το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit. Σα ευχαριστώ για την ερώτησή σα ε, για το Ηνωμένο Βασίλειο και για το Brexit. Ε. Εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο εξ ονόματος της ε, τομέα της ναυτιλίας. Πολύ φοβάμαι ότι και πάλι θα χρειαστεί να επαναλάβω αυτά που είπα. Όλα αυτά εξαρτώνται από το πώς θα δημορφωθεί η εμπορική συμφωνία. Τι θα συμφωνηθεί τελικά. Αν υπάρχει μεγάλη διαφορά με την τρέχουσα κατάσταση, δεν θα υπάρχει μειονέκτημα, αλλά αυτά που ακούμε από τον Μπαρνιέ για παράδειγμα, δεν ε, μας υποδεικνύουν ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Θα αλλάξουν τα πράγματα και όχι προς τη θετική κατεύθυνση. Αυτό δεν θα είναι καλό ούτε για το Βασίλειο, ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι οι ενδείξεις που έχουμε ακόμα. Ανησυχούμε λοιπόν, ανησυχούμε και ενδεχομένως να αποτελεί πολιτικό μήνυμα αυτό το οποίο ακούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εμείς αυτό το μήνυμα λαμβάνουμε διαρκώς. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι στην τελική ανάλυση κατά πόσον τελικά θα καταλήξουμε σε μια χειρότερη κατάσταση από αυτή που ξέρουμε και γνωρίζουμε. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό το οποίο μας απασχολεί ως κλάδο. Κύριε Ρικέ, χρειαζόσαστε περισσότερο από ένα λεπτό. Μα ποια θα είναι τα ευεργετήματα. Ακούω τις ανησυχίες σας, αλλά πιστεύετε ενδεχομένως ε, να υπάρχουν και θετικά. Μετά το Brexit για το Ηνωμένο Βασίλειο πάντα. Κοιτάξτε, αυτό που ενδεχομένω να συμβεί και το είπα και εισαγωγικά είναι το εξή. Α υποθέσουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα βελτιώσει το επιχειρηματικό του κλίμα σε σχέση με την Ευρώπη και έτσι θα δημιουργηθεί διαγωνιστικό πλεονέκτημα. Τότε ενδεχομένω οι ευρωπαϊκέ εταιρείε, οι ναυτιλιακέ, να αναλογιστούν, να φτιάξουν υποκατάστημα στην, ε, στον Εμένο Βασίλειο να επεκτείνουν το υποκατάστημα που έχουν. Και αυτό φυσικά θα πρέπει να προσέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα συμβεί τελικά στην Βρετανία, θα έχουν δυνατότητε να το κάνουν αυτό, θα το χρησιμοποιήσουν, θα το εκμεταλλευτούν αυτό. Και αυτό μπορεί να συμβεί. From the perspective... Από πλευρά ε, ταξιδιών αναψύχη, εμεί είμαστε το δεύτερο μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρώπης, αλλά μόνο 4% του δικού μας πληθυσμού αγοράζει ταξίδια αναψυχής. Γι' αυτό θα πρέπει να αναπτύξουμε την ε, ντόπια αγορά. Θεωρούμε ότι έχουμε να κάνουμε με την τρέχουσα κατάσταση που δεν αλλάζει. Business as usual. Νομίζω ότι από πλευράς P&O Ferries θα μπορέσουμε να μετασχηματίσουμε τις υπηρεσίες μας και να το κάνουμε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αν δεν είχαμε Brexit. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κλούνη για τρία λεπτά. Ε, σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τους ομιλητές για τις εισηγήσεις τους. Ε, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο θέμα, δεν υπάρχει βεβαιότητα και έτσι δεν μπορούμε να προβλέψουμε τίποτα. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι η κυβέρνηση του ε, Ηνωμένου Βασιλείου είπαν ότι δεν θα συμμετέχουν ε, ούτε στην εσωτερική αγορά ούτε στην Τελωνιακή Ένωση. Ε, όσον αφορά το θέμα της τεχνολογίας, κυρία Μακένζη, το οποίο αναφέρατε αρκετές φορές και νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό και ε, κύριε Ντόρφμαν, αναφερθήκατε στην ομαλή χωρί τριβέ ε, θαλάσσια ε, ε, ναυτιλία. Πιστεύετε ότι η τεχνολογία μπορεί να προβλέψει κάτι τέτοιο. Ε, συμφωνώ απολύτως με τις παρατηρήσεις ότι η τεχνολογία μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και σε περίπτωση που μπορεί να υπάρξουν ε, επιπλέον απαιτήσει για τους ε, επιβάτες. Ε, για παράδειγμα, εάν πρέπει να συμπληρώσουν κάποιο έντυπο, μπορεί να το κάνουν αυτό από το σπίτι τους, από τον υπολογιστή. Συμφωνώ απολύτως ότι η τεχνολογία μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Κυρία Μακένζη, ναι, συμφωνώ και εγώ απολύτως. Αν δούμε πόσο έχει οθετήσει νέες τεχνολογίες ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι διαπιστώνουμε αυτό και είναι ευκαιρία να εξετάσουμε τις νέες τεχνολογίες, τεχνολογίες που ήδη υπάρχουν, να τις χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο και για να βελτιώσουμε ε, την ε, εμπειρία των καταναλωτών, ε, των πελατών, των μας, αλλά και για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του Brexit. Ε, όσον αφορά την ενιαία αγορά ναυτιλίας, Πιστεύετε ότι δεν υπάρχει έτσι, δεν είναι, ότι υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις σε όλη την ε, Ευρώπη, διαφορετικοί κανόνες. Αυτό δεν είναι κάτι που σχετίζεται με το Brexit, αλλά είναι σημαντικό θέμα για την αυτιλία. Νομίζω ότι αναφέρεστε Ε, στην οδηγία για τις ε, διατυπώσεις, ε, τι πρέπει να κάνει κανείς για να μπει σε ένα λιμένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγματι, αυτό αποτελεί σημαντική πρόκληση για τα πληρώματα των σκαφών αυτή τη στιγμή. ελπίζουμε σύντομα να λάβουμε, το, το συντομότερο δυνατό να λάβουμε πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διεκπαιρεώσει ε, σύντομα το θέμα. Είναι όμως ε, θέμα το οποίο θα πρέπει να λύσει η πολιτική. Συμφωνώ με αυτό που λέτε, αλλά φυσικά όλα αυτά συνεπάγονται και κάποιο κόστος και για τις μικρές ε, επιχειρήσεις, για τους μικρούς εφοπλιστές ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα των διατυπώσεων. Ναι, η απάντηση είναι η τεχνολογία, ε, συνεπάγεται όμως και κάποιο κόστος. Ναι, ήθελα να δω τι μπορεί να γίνει από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για να γίνουν πιο αποτελεσματικοί οι λιμένες. Έχει τελειώσει ο χρόνος μου, αλλά θα ήθελα απλά να πω ότι ελπίζω ότι θα είναι πάντα ευπρόσδεκτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ναυτικοί και οι επιβάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, ε, άλλωστε στην ε, Ιρλανδία είναι οι πιο τακτική μας επισκέπτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κλούν. Κύριε Κιστελεφ, επανήλθατε και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πολύ καλή η ερώτηση. Ποια θα είναι τα ευεργετήματα μετά το Brexit και θα υπάρχουν. Νομίζω. Νομίζω ότι το πάνελ μας είπε ότι όχι. Γιατί η Βρετανική κυβέρνηση λέει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Τελωνιακή Ένωση. Δεν βλέπω να μην υπάρχουν επιπτώσεις στις θαλάσσιες μεταφορές, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αγαθά. Δεν περιμένω απάντηση, αλλά ε, θα ήθελα να ρωτήσω το πάνελ, θα ευεργετηθεί η Ευρώπη εάν ευεργετηθεί από το Brexit. Νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να αναθεωρήσουμε τα πάντα και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δράσουμε στο μέλλον. Νομίζω ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να προβούν σε επαναδιαπραγματεύσεις και όλοι θα ευεργετηθούμε κατά κάποιο τρόπο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Τέιλορ. Και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να προτρέξω σε αυτά που είπατε κύριε Ντόρφμαν. Ας δούμε το χειρότερο σενάριο. Εάν δεν επέλθει η συμφωνία, τότε θα πρέπει να καταβληθούν δύο φορές ε, οι δασμοί για να μπουν αγαθά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το έχετε προβλέψει αν δεν επέλθει η συμφωνία καταβολή διπλών δασμών δηλαδή. Αν δεν επέλθει συμφωνία, θα ισχύσουν οι κανόνες του ΠΟΕ, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Και μπορούμε λοιπόν να επιβάλλουμε ε, δασμούς και το καθεξής. Ε, δασμοί οι οποίοι έχουν μειωθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Αλλά η κατάσταση θα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που είναι τώρα. Και ενδεχομένως, ναι, να επιβληθούν τέτοια τέλη. Αλλά επαναλαμβάνονται ότι αυτό εξαρτάται από το πώς θα τελικά η κατάσταση. Η θέση μας είναι σαφής. Ε, πάντα θα υπάρχει αμφίδρομη κίνηση και θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια υποστηρικτική υπηρεσία με τη χρήση της ε, υψηλής τεχνολογίας. Δεύτερη ερώτηση. Κατά πόσο το Brexit μπορεί να αλλάξει τον δελεαστικό χαρακτήρα ορισμένων γραμμών. Ξέρουμε ότι υπάρχουν εταιρείε που κάνουν εισαγωγές, εξαγωγές, λιμάνια με συγχωρείτε. Υπάρχουν δηλαδή λιμένες εισαγωγών, εξαγωγών. Εάν προσθεθούν σύνορα υπάρχει ευεργέτημα και επίσης τα υπηρετικά λιμάνια Άμστερνταμ, Ρότ, Ρότερνταμ, Ζέμπρουγκε θα μπορέσουν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους με βάση αυτά τα νέα δεδομένα. Αυτό το έχετε σκεφτεί. Δεν έχουμε κάνει σχετική μελέτη για την μετατόπιση των εμπορικών ροών, οι οποίες δεν ενδεχομένω να προκύψουν. Μια γενική παρατήρηση όμως ότι αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα, και το κοιτώντα για παράδειγμα το τι κάνει η Κίνα που επενδύει στον Πειραιά. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση και στο ρόλο που Και αυτά πάντα υπάρχουν στην δυνατότητα. Ένα νέο σύνορο, αν μπει και το πώς θα δημορφωθεί, Αυτό είναι κάτι το οποίο πάντα θα κοιτάνε οι μεταφορείς και το πώς θα αντιμετωπίσουν τέτοιες ε, αλλαγές των διαδρομών. Αυτά θα επηρεάσουν τις συζητήσει μας ε, εδώ στο Κοινοβούλιο για την Αυτιλία και για το ETS. μπορεί ενδεχομένω το Ηνωμένο Βασίλειο να καταστεί ξαφνικά πάρα πολύ ελκυστικό για την Κίνα Ω ε, σημείο κοντινό προ την υπηρετική Ευρώπη σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το ETS. Ε βλέπουμε λοιπόν μια σειρά ε, θεμάτων που μπορεί να επηρεάσουν του το πώς θα διαμορφωθούν οι εμπορικές ροές και πώς θα μετατοπιστούν. Αυτό εξαρτάται και από τα σύμφωνα και από τις συμφωνίες και το πώς τελικά θα καταφέρουμε να προσαρμοστούμε στην κατάσταση. Μάλιστα, να δώσω το λόγο στην κυρία Άντερσον και στον κύριο Φαντεκάμ για να κλείσει. Για να υποστηρίξω αυτά που είπε ο κύριος Ρεκέ για το θέμα της ανάπτυξης επιχειρήσεων τα τελευταία δέκα χρόνια είδαμε απώλεια διαδρόμων για τους επιβάτες μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Σκανδιναβίας. Εγώ αυτό που φοβάμαι ότι είναι ότι και άλλες διαδρομές θα περιοριστούν πολύ απλά γιατί υπάρχει αβεβαιότητα. Για παράδειγμα, από το Κόρκ βλέπω ότι υπάρχει φέρει προς την Ισπανία από φεύγοντας το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό δεν ε, είναι μια ανησυχία ότι δηλαδή ο κλάδο ολόκληρο θα προσπαθήσει να αποφύγει το Ηνωμένο Βασίλειο όπου αυτό είναι δυνατόν. Απάντηση. Αυτό κάπω συνάδει με αυτά που είπα στην τελευταία μου απάντηση ότι αν αλλάξουν τα πράγματα ασφαλώ η βιομηχανία, ο κλάδο, μάλλον θα ψάξει να βρει τι απαντήσει που χρειάζεται. Αυτό ενδεχομένω είναι μια πραγματική συνέπεια. Ο κλάδος θα ψάξει να βρει επιχειρηματικέ λύσει εκτός μικροφώνου. Ναι, συγγνώμη. Οι εταιρείε πάντα ψάχνουν νέες, ε, νέους Αυτό δεν έχει αλλάξει προφανώς ενώπιση του Brexit. Και νομίζω ότι από πλευράς ε, κρουαζιέρας ο προορισμός είναι αυτός που μετράει. Όπου θέλει να πάει ο κόσμος και εφόσον είναι εύκολο να το πετύχουμε αυτό το προορισμό. Ο κ. φοντενκάμπ για να κλείσει τη συζήτηση. Α, μάλιστα, λέει ο κ. Ε, φοντενκάμπ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω όλους ε, τους συμμετέχοντες από πλευρά του κυρίου Πίπερ. Έχω μία ερώτηση να κάνω. Ωστόσο, στην εισαγωγή του κυρίου Ντόρσμαν άκουσα τη λέξη offshore, την είπατε. Δεν μπορούσα να μας πείτε δύο λόγια εδώ, γιατί μιλάμε εδώ για υφαλοκρηπίδες υπηρετικές υφυλοκρηπίδες, οι οποίες ε, είναι κοντά η μία στην άλλη. Αναμένεται προβλήματα εφοδιασμού, ερμηνείας ε, των κανόνων. Γιατί δεν αναφέρετε το θέμα αυτό, γιατί δεν είπατε αυτή την έκλεξη, τη λέξη. Έχει να κάνει με την πρόσβαση στην αγορά. Για μεταφορά επίσης ε, ως υπηρεσία εξυπηρετική του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Υπάρχει λοιπόν το θέμα του εφοδιασμού τέτοιων ε, τοποθεσιών σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τη μεταφορά προσωπικού, τροφίμων, εγκατάσταση ανεμόμυλων. Φυσικά πάντα υπήρχε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Τώρα έχουν προσταθεί και οι ανεμογεννήτριες. Θα έχουμε και άλλες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Είναι θέμα πρόσβαση στην αγορά. Οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πρόσβαση στη Βρετανία και αντίστροφα. Είναι εντελώς ανοιχτή η κατάσταση. Αυτό ανησυχούμε. Αυτό μας ανησυχεί. Δεν πρέπει να αλλάξει αυτό. Να θέσει, για παράδειγμα, απαιτήσει το Ενωμένο Βασίλειο για τις σημαίες, για το προσωπικό, για τους υπαλλήλους. Αν αρχίσει το Ενωμένο Βασίλειο να φέρει τέτοιες ε, απαιτήσει. Κοιτώντα τι γίνεται στην Αμερική, καταλαβαίνουμε όλοι τι συμβαίνει, αλλά δεν θέλουμε να συμβεί προφανώ το ίδιο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό μα απασχολεί και αυτό ζητούμε να το προσέξετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Ευχαριστώ, λέει και πρόεδρο. Ευχαριστώ το πρώτο πάνελ και νομίζω ότι μπορούμε να σας χειροκροτήσουμε κύριε Ντόρσμανς, κύριε Γκρίφιτς και κυρία Μακένζη, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που μας ε, παρουσιάσατε κάποια ζητήματα τα οποία καλούμαστε να τα σκεφτούμε και όλοι συμφωνούμε σε ό,τι αφορά την ανάγκη να υπάρχει αυτή η μεταβατική περίοδος, να προσαρμοστούμε, να έχουμε δυνατότητα να προσαρμοστούμε, όποιοι και αν είναι οι κανόνες. Αλλά προφανώς δεν γίνεται σε μία νύχτα να υλοποιηθεί μία συμφωνία. Χρειάζεται μεταβατική περίοδος. Το ακούσαμε λοιπόν και θα καταλάβουν ό,τι μπορούν να καταλάβουν ε, οι διαπραγματευτέ, αλλά μπορείτε να υπολογίσετε στην ε, Επιτροπή Μεταφορών για τι θα προασπιστεί τα δικαιώματά σα. Και τώρα να περάσουμε στο δεύτερο πάνελ. nous continuons. Je vais demander à... Θα ήθελα ο κύριος Ζωακίμ ε, Κοέν, η ε, rejoindre Ζωακίμ Κοέν, Λάιτον. Να έρθουν εδώ. Ευχαριστώ για τους, τους τρεις ομιλητές που δέχτηκαν την πρόσκλησή μας. Θα περάσουμε λοιπόν τώρα στους λιμένες. Θα αρχίσουμε με τον κύριο Κουένς, μια και είμαστε στο Βέλιο. Σας ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Είσαστε διευθυντής του λιμανιού της Μπρούζ και θα μας ε, κάνετε μια παρουσίαση για τις συνέπειες του Brexit σε σχέση με το λιμάνι σας. Έχετε το λόγο για 7 λεπτά και μετά θα συζητήσουμε το θέμα. Κύριε Κοένης, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι κυρίε και κύριοι και στι τρει γλώσσε. Ε, ε, ο κύριο Κούντ. Μιλάμε για το εμπόριο, εμπόριο και λιμένε. Κοιτάξτε στο μπρου τι γίνεται, είναι, είχαν σε αττικές ε, πόλεις του 14ου αιώνα με εμπόριο προ το Ηνωμένο Βασίλειο. Από το 14ο αιώνα λοιπόν υπάρχει αυτό το εμπόριο και θα συνεχίσει να υπάρχει εμπόριο και του επερχόμενου αιώνε με ή χωρίς Brexit θα έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε για την ε, μεταφορά ε, εμπορευμάτων προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Ιδιαίτερα σήμερα βρισκόμαστε εδώ, γιατί πιστεύω ότι η θέση μας είναι σαφέστατη σε ό,τι αφορά το εμπόριο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φέρνουμε αγαθά από όλη την Ευρώπη. Τα μεταφέρουμε με διαοδού, δια και διαθαλάσσεις ε, προς τις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, τη Σκανδιναβία και τη Ρωσία. Για μα, λοιπόν η ευρωπαϊκή αγορά είναι σημαντική. 46% της ευρωπαϊκού εμπορίου προορίζεται προ το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι μεταφέρουμε ε, εμπορεύματα από όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και προ την Ηνωμένο Βασίλειο. Κοιτώντας ε, τα προϊόντα τα οποία παράγονται κυρίως στη Βόρεια Γαλλία, στο Βέλγιο, κοντά στους λιμένες, φαντουργικά προϊόντα. Έχουμε μεγάλο τομέα της μηχανίας, τρόφιμα, α, αυτοκίνητα και εξαρτήματα, φαρμακευτομιομηχανία, όλα αυτά εξαγάγονται προς το Ηνωμένο Βασίλειο. 67% όλου του εμπορίου μας είναι Εξαγωγέ και μόνο το υπόλοιπο είναι εισαγωγέ από όλη την Ευρώπη, από την Ανατολική Ευρώπη, Ρουμανία, Ουγγαρία και από την Ιταλία. 53 τρένα κάθε εβδομάδα από την Ιταλία προ το Ζεμπρίχε που μεταφέρουν αγαθά μεταξύ άλλων και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Εστιαζόμαστε λοιπόν σε ιστορικού συνδέσμου, αλλά και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Από πλευρά Ηνωμένου Βασίλειου, κοιτάξτε, στο Λονδίνο μέχρι και τον Βορρά μεταφέρουμε αγαθά. Είναι ένας πολύ εξατομικευμένος τρόπος μεταφορών με εμπορεύματα τα οποία δεν έχουν, δεν συνοδεύονται. Και έχουμε 5.000 ε, άμεσες θέσεις εργασίας που συνδέονται με το εμπόριο αυτό. Το σημαντικό είναι τα προϊόντα, οι βιομηχανίες. Έχουμε 70 μεταφορές κάθε εβδομάδα. Το πρόβλημα είναι τη μεταφορά των εμπορευμάτων στους λιμένες. Ε, έχουμε 2.000 άτομα που ασχολούνται μόνο στις αποθήκες απασχολούνται. Την επόμενη μέρα είναι στο Λανδίνο, στο Μπερμίγκαν, στη Γλασκόβη ή όπου τα χρειάζονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να είναι πολύ στην ώρα της πάντα οι υπηρεσίε μας. Είναι ιδιαίτερα φυσικά για τα τρόφιμα και για άλλα προϊόντα που χαλάνε. Επίσης και ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι πολύ σημαντικός. Είμαστε παγκόσμιο ηγέτης σε αυτοκίνητα, παραγωγή αυτοκινήτων. Από τη Γερμανία, από τη Γαλλία προς τον Βασίλειο μεταφέρουμε εξαρτήματα, αλλά και από την Απανατολή, από το Μεξικό και από τις ΗΠΑ. Περίπου 8 δις, 1 δις εκατομμύριο περίπου αυτοκίνητα. 70% είναι η προσεξαγωγή και πολύ σημαντικό αυτό φυσικά για τη μηχανία και για τους λιμένες. Και για τον Εμένα Βασίλη είναι σημαντικό αυτό το εμπόριο. Αυτό τι σημαίνει ότι πολλά από τα αγαθά αυτά είναι σε διαμετακόμιση περνούν από την Ευρώπη. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν λοιπόν αυτές οι επιχειρήσεις όπως το Toyota που έχει μια εταιρεία βάση, με βάση στο λιμάνι μας και θέλει να λαμβάνει προϊόντα όχι μόνο από τη Βαλενσιana, από την Βορειοκαλία, αλλά και από την Ιαπωνία, την Νότια Αφρική, από την Τουρκία, μέσω των λιμένων. Πάρα πολλέ ιδέες εργασίας. Να δούμε και το Brexit έχει ληφθεί η απόφαση για το Brexit. Τι θέλουμε. Θέλουμε μια συμφωνία εμπορική, γιατί ήδη σήμερα αντιμετωπίζουμε τις ε, δυσκολίες ε, σε ό,τι αφορά την ισοτιμία μεταξύ λίρας και ευρώ. Γιατί υπάρχει ανταγωνισμός με χώρες εκτός Ευρώπης, όπως με την Τουρκία για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την κλωστοφαντουργία. Έτσι έχουν τα πράγματα. Αν σε όλα αυτά λοιπόν προσταθεί και το σενάριο των ε, προδιαγραφών του ΠΟΕ δασμού 10% για παράδειγμα για φρούτα, σοκολάτες. Δεν ότι αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Μία χώρα όπως το Βέλγιο θα πλήρωνε 1,6 δις ευρώ για τέτοιους τελωνιακούς δασμούς και θα λάμβανε φυσικά και ε, έσοδα από τους δασμούς, αλλά πολύ λιγότερους. Ε, μία στις 40 λοιπόν δουλειές στη Φλάνδρα έχει να κάνει με τη μεταφορά προϊόντων και θα είχαμε πολύ σημαντικές. Πώς μπορούμε λοιπόν να προετοιμαστούμε, τι κάνουμε. Έχουμε ακούσει πολλές ερωτήσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις τελωνιακές ε, διαδικασίες. 47% υπολογίζεται ότι θα αυξηθούν αυτές οι εκτελονίσεις. Και οι λιμενικές αρχές ε, καταρτίζουν ένα ψηφιακό σύστημα για την σύνδεση όλων των δεδομένων. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωφέλιμο και χρήσιμο αν θα μπορούσαμε να είχαμε υποστήριξη από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις τελωνιακές υπηρεσίες από την υπηρετική Ευρώπη, για να ξεκινήσει αυτή η πλατφόρμα. Επίσης σημαντικό είναι να υπάρχουν διαπραγματεύσεις και με τους άλλους λιμένες από την άλλη πλευρά. Και τέλος, θα πρέπει να υπάρχει και μια σαφή μεταβατική περίοδος. Το είπαμε ήδη σήμερα. Θα πρέπει να υπάρξει μία αλλαγή μετά τη μεταβατική περίοδο, όχι στη φάση τη μεταβατική και μετά τη μεταβατική αυτή φάση. Καλό θα υπάρχει μία μόνο φάση αλλαγής. σαφήνια προφανώς χρειάζονται, σαφής εμπορική συμφωνία για να αντιτηρηθεί η ελεύθερη μετακίνηση αγαθών και σε ό,τι αφορά τα διεθνή εμπορεύματα που περνούν από τα βελγικά λιμάνια, τα ευρωπαϊκά λιμάνια και φυσικά είναι σημαντικά όλα τα στοιχεία αυτό που θα θέλαμε είναι το συντομότερο δυνατό να, ξεκινήσουν να ξεκινήσουν οι προετοιμασίε που να μην περιμένουμε μέχρι το τέλο των διαπραγματεύσεων για να ξεκινήσει η προσαρμογή και φυσικά έχουμε και κάποια θέση σε ό,τι αφορά τους ίδιου όρους ανταγωνισμού. Θέλουμε να αποφύγουμε τις διμερείς συμφωνίες. Θα πρέπει να βρεθούμε στην ίδια θέση με τις άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες. Και φυσικά χρειάζεται πιο πολύ διάλογο για το εμπόριο με την Ιρλανδία. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Monsieur Ευχαριστούμε κύριε Κοέν για αυτή την παρέμβαση και τηρήσατε και το χρόνο σας. Επιμείνατε για την ε, περίοδο ε, μετάβασης αλλά και σαφήνεια των κανόνων. Δίνω το λόγο σε εσάς κύριε Ράιλι από το λιμάνι του Δουβλίνου και έχετε να μας κάνετε και μια παρουσίαση. Έχετε το λόγο. Um, I'm Ευχαριστώ. Από τον λιμένα του Δουβλίνου έρχομαι, που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ιρλανδίας. Είμαι μηχανικός και η πρόκλησή μας εκεί είναι η δημιουργία υποδομών ε, πρέπει να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα και το Brexit δημιουργεί τεράστια βεβαιότητα για μας, κάτι πολύ ε, προβληματικό όταν θέλει κανείς να κάνει σχέδια για το μέλλον. Θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω στις πέντε ερωτήσεις που μας τέθηκαν. Τον Δεκέμβριο άρχισαν κάπως να γίνονται πιο σαφή τα πράγματα που ο κύριος ε, Μπαρνιέ ε, παρουσίασε τη διαφάνεια που βλέπετε που δείχνει τις διάφορες επιλογές μετά το Brexit και συγκρίνοντάς τες με, την, ε, με τις κόκκινες γραμμές των Βρετανών. Εμείς πιστεύουμε ότι το Brexit είναι Brexit, οπότε δεν έχει σημασία αν είναι σκληρό ή ήπιο. Ε, δεν έχουμε εναλλακτική λύση. Πολιτικά ε, είναι άλλη ιστορία. Όπως όμως ε, υπόθηκε νωρίτερα, πρέπει να ελπίζουμε για το καλύτερο, αλλά να προετοιμαστούμε για το χειρότερο. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε σχέδια όσον αφορά την υποδομή του λιμένα. Και έχοντας αυτό κατά νου, ξεκινήσαμε τον σχεδιασμό το, της υποδομής ε, για τους ε, σταθμούς διέλευση των συνόρων στο λίμενα του Δουβλίνου. Αυτό δεν είναι ε, καμιά πάρα πολύ δύσκολη επιστήμη, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα τελωνία και την αστυνομία και τη συνοριοφυλακή κλπ. Ε, μέχρι τον ε, Δεκέμβριο θα έχουμε έτοιμα τα σχέδια μας, κατόπιν ε, θα λάβουμε την σχετική άδεια και σκοπεύουμε να τα έχουμε όλα έτοιμα τον Μάρτιο του 2019. Εάν δεν χρειαστούν, τόσο το καλύτερο. Αλλά καλύτερο να έχουμε την υποδομή και ας μην χρειαστεί παρά να μην την έχουμε και να χρειαστεί. Όσον αφορά τα αριθμητικά στοιχεία, τι σημαίνει το Brexit για την Ιρλανδία. Ε, ο κύριος Δόσμαν μας έδωσε κάποια δεδομένα. Ε, το Δουβλίνο ήδη δέχεται πλοία από εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπου 2.000 ε, μονάδες φορτίων το χρόνο. Και μέσα σε μία νυχτή θα αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός αυτός και με βάση αυτό θα πρέπει να σχεδιάσουμε το μέλλον. Μετά το Brexit το Δουβλίνο θα παραμείνει το μεγαλύτερο λιμάνι για το, την Ιρλανδία με το 88% των ferry boat, των οχηματογωγών ρο-ρο. Ε, πολλά από αυτά τα πλοία πηγαίνουν ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λίβερπουλ κλπ. Αλλά και πολλά πηγαίνουν ε, σε ευρωπαϊκά λιμάνια. Εδώ βλέπετε το μεγαλύτερο οχηματογωγό ε, του κόσμου τέτοιου τύπου. Λέγεται ε, Σελήν από το Ρότερνταμ ε, και έχει τεράστια χορηκτικότητα και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μας χρησιμοποιεί τώρα αυτό το πλοίο από το Schleswig-Holstein από τα ναυπηγεία εκεί και τον, φέτος τον Μάιο θα αρχίσει οι διαδρομές προς το Χερβούργο. Εάν ακολουθηθεί αυτή η τάση, διότι και η Irish έχει ανακοινώσει το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλιο του κόσμου, ε, αλλά αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ ευέλικτος ο τομέας και βλέπουμε ήδη πολλές διαδρομές κατευθείαν από το Δουβλίνο στην υπηρετική Ευρώπη και πιστεύουμε ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί. Ε, είναι πολύ ψηλά τα γράμματα στις ε, διαφάνειες, ε, ούτε εγώ δεν μπορώ να τα διαβάσω, θα πρέπει να θυμηθώ τι έγραφα. Μας ερώτησαν σχετικά με πιθανές αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο μετά το Brexit. Ουσιαστικά θα έχουμε πενταπλάσια αύξηση του αριθμού των φορτίων που θα χρειάζονται εκτελονισμό. Ε, θα ε, έχουν την ίδια μεταχείριση οι Βρετανοί με τους Κινέζους ε, και γι' αυτό το ενδεχόμενο ετοιμαζόμαστε. Θα έχουμε αύξηση του τομέα λειτουργικής υποστήριξης και νομίζω ότι θα έχουμε αντιστροφή αυτού που είδαμε το 1985, ε, όπου είχαμε μεγάλη απλοποίηση και μείωση του κόστους. Μας ρώτησαν πώς ε, επηρεάζει το Brexit ε, τα σχέδια μας για τα επόμενα 5-10 χρόνια. Σχεδόν καθόλου προβλέπεται να αυξηθεί κατά 17% ο πληθυσμός της Ιλλανδίας μέχρι το 2040. Οι όγκοι λοιπόν θα αυξηθούν πολύ, ενώ οι προκλήσεις του Brexit είναι τόσο ε, βραχυπρόθεσμες που δεν επηρεάζουν την, ε, τον προγραμματισμό για την υποδομή στον λιμένα του Δουβλίνου. Θα προσπεράσω πολύ γρήγορα τις επόμενες ε, δύο διαφάνειες. Το μόνο που λέω εδώ είναι ότι είναι μεγάλη πρόκληση το Δουβλίνο να γίνει ένας από τους κεντρικούς λιμένες ε, του δικτύου, των διευρωπαϊκών δικτύων TNT. Ε, σε 57 εβδομάδες όμως ε, θα ζήσουμε την πραγματικότητα του Brexit. Γενικά αργό πολύ να υιοθετήσω νέες διαδικασίες και τεχνολογίες μέσα σε 57 εβδομάδες δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι ρεαλιστικό. Να επανέλθω στην ε, παρατήρηση της κυρίας Μακένζη. Εμένα με ανησυχεί κάπως ότι διάφορες επιχειρήσεις πιστεύουν ότι όλα θα συμβούν από μόνο τους ε, χωρίς να χρειαστεί δράση ε, από καμία πλευρά. Θα χρειαστεί δράση από πλευράς των λιμένων όσον αφορά τις υποδομές, από τους μεταφορείς, από τις εταιρείες οχηματογωγών θα πρέπει όλοι αυτοί να συμμορφωθούν με τις τελωνιακές ρυθμίσεις του Ενωσιακού Τελωνιακού Κώδικα. Και για μένα είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αυτό είναι το σενάριο με βάση το οποίο εργαζόμαστε. Μία από τις ερωτήσεις ήταν τι μήνυμα έχουμε προς τους διαπραγματευτές. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού μας ε, έχουμε ξεκινήσει διάλογο σχετικά με ε, την δυτική ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου και ε, μία από τις επαφές μου εκεί μου είπαν ε, ότι το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι δεν έχουμε σαφή απάντηση από πλευράς της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Εγώ αυτό που θα ρωτούσα τους διαπραγματευτές θα ήταν πέρα από το να έχουμε απολύτως ομαλή μετάβαση στο μέλλον να φροντίσουμε οι Βρετανικοί λιμένες να είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Και φυσικά πάντα πιστεύουμε να μην δούμε τις χειρότερες, ε, τις ε, χειρότερες συνθήκες, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι αν ζήσουμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Λάιτον για 7 λεπτά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν ε, έχω γραφικές ε, παραστάσεις μαζί μου. Ονομάζομαι David Layton, είμαι επικεφαλής των εταιρικών υποθέσεων στα Βρετανικά λιμάνια. Θα ήθελα να σταθώ σε τρία σημεία. Καταρχήν η εισήγηση για το εμπόριο που διαχειριζόμαστε με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός. Δεύτερον, οι, τις επιπτώσεις ε, ε, του Brexit στα Βρετανικά λιμάνια και τέλος ε, τις ε, ενδεχόμενες επιπτάσεις. Η ABP είναι ο, η μεγαλύτερη επιχείρηση λιμένων στο ε, ε, Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε 21 λιμάνια στην Αγγλία, ε, Σκοτία, Ιρλανδία και Ουαλία. Έχουμε 119.000 θέσεις εργασίας και συνεισφέρουμε κατά 70 δις στερλίνες ετησίως. Το αυτό του εμπορίου μας σχετίζεται με κράτη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 55 με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η κατανομή διαφέρει. Όταν δούμε ε, με μονομένες, ε, μονομένες λιμένες, δηλαδή εμείς δρούμε στο Southampton όπου υπάρχουν εμπορευματοκιβώτια ταξίδια αναψυχής, εμπόριο και το 36%, το, τα 36 δις τερλινών αφορούν το εξωτερικό εμπόριο, δηλαδή χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέσσερις ε, ε λιμένες στην Ανατολική Αγγλία έχουν ένα 60% του εμπορίου με το ε, με τις ευρωπαϊκές χώρες. Πέρσι είχαμε 665.000 ε, ε, μεταφορές με τρέλερ και μεταφορές ρορό. Και επίσης είχαμε και ασυνόδευτες ρορό αποστολές. Επίσης, 345.000 ε, εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στα λιμάνια από το Brexit. Ας υποθέσουμε ότι θα ε, αποχωρήσουμε από την Τελωνιακή Ένωση. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για την οικονομική μας ανάπτυξη, βράχη και μακροπρόθεσμα θεωρώ ότι ο συνολικός ε, αριθμός, ε, ο όγκος του εμπορίου θα εξαρτηθεί από το μελλοντικό εμπόριο. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για τα υπέρ και τα κατά, απλώς θα ήθελα να μιλήσω για τις επιπτώσεις, για τις ε, εμπορευματομεταφορές. Όλα εξαρτώνται από λιμάνι σε λιμάνι δηλαδή σε σχέση με εμπόριο εντός και, Ευρω... και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας ενδιαφέρουν δηλαδή οι λιμένες ε, που έχουν μεταφορές ρο-ρο προς και από την Ευρώπη. Ε, ίσως χρειάζονται επιπρόσθετες, ε, επιπρόσθετη τελωνιακή έλεγχη που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα ιδιαίτερα εκεί που δεν υπάρχει χώρος. και ίσως υπάρξουν ενδεχόμενες καθυστερήσεις στο Ντόβερ. και αυτό μας απασχολεί και ιδιαίτερα πρόθεσμα. Υπάρχει κίνδυνος καθυστερήσεων, ιδιαίτερα στο Ντόβερ και θα δούμε τι θα γίνει με το κάργο που εισέρχεται εκτός από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέες τεχνολογίες μας δείχνουν ότι ένα μόνο ένα 1,3% μεταφορών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σταματάει για ελέγχους, ιδιαίτερα για λόγους υγείας, για την ασφάλεια των τροφίμων. Άρα, την ε, πρώτη μέρα αποχώρησης, η ρυθμιστική ε, οι ρυθμίσεις ορίζουν να γίνονται έλεγχοι ιδίω για λόγους υγείας και υγιεινής, ε, κρέας, πουλερικά και ούτω καθεξής. Άρα, δεν χρειάζονται περισσότεροι έλεγχοι όταν θα είμαστε εκτός τελωνιακής ένωσης. Φαίνεται λοιπόν ότι οι έλεγχοι δεν θα αυξηθούν σε σημείο ώστε να διαραγεί το εμπόριο. Ως προς το, τις μεταφορές ρορό και ιδιαίτερα στο ντόβερ, εάν γίνουν καθυστερήσεις, δεν θα είναι απότοκες ε, ε, αυτών των νέων παραγόντων και θεωρώ ότι όλα εξαρτάται εξαρτώνται από το πώς η πολιτική σκέψη θα ε, διέπει τις σχέσεις και από τις δύο πλευρές. Εάν λοιπόν υπάρχει μία μεταβατική περίοδος, τότε θα αρχίσουμε να αναπτύσσουμε αυτά τα συστήματα ε, τώρα για να αποφύγουμε τα προβλήματα. Μιλώντας όμως για τις επιπτώσεις του ε, Brexit, μπορεί να υπάρχει μία ε, συγκεκριμένη δυσχέρανση μεταφορών ρόρο. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα εμπορευματοκιβώτια και τα, τις ασυνόδευτες ρόρο μεταφορές. Και αυτό αφορά και τη μεταφορά εμπορευμάτων. Θα ήθελα να πω ότι Συνεργαζόμαστε με τα λιμάνια, όλα τα λιμάνια στην Ευρώπη για την ε, ABP. Έχει μεγάλη σημασία να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες για τους πελάτες μας και όλοι θεωρούν στη Μεγάλη Βρετανία ότι θα πρέπει οι κινήσεις εμπορευμάτων να παραμείνουν και να κινούνται απρόσκοπτα. Οι Ευρωπαίοι είναι φίλοι μας και εταίροι και θεωρούμε ότι θα συνεχίσουμε την ε, ανωδική πορεία της ε, ανταλλαγής εμπορευμάτων. Λοιπόν, άρχεται η συζήτηση. Διαδικασία πινκ-πονγκ, λοιπόν, για πέντε λεπτά δίνω το λόγο στον κύριο Βίμ Βαντεκαμ. Να παρακαλώ όσοι θέλουν το λόγο να το ρωτήσουν τώρα. Κύριε Άντερσον. Allez-y, θα ήθελα να πω ευθύς εξ αρχής ότι εδώ στο Κοινοβούλιο μια πολύ μικρή ομάδα πολιτικών, μια πολύ περιορισμένη ομάδα πιστεύει ότι είναι αδύνατο να γίνει το Brexit. Και ξέρετε ότι και εγώ συγκαταλέγομαι στην ομάδα αυτή, το λέω να ακουστεί και σήμερα το απόγευμα. Να συνεχίσουμε τον κύριο Κούντσο Μία παρατήρηση πιο πολύ. Γιατί είμαι εγωιτευμένο και εντυπωσιασμένο από την, από την παρατήρησή σα θέλετε μία μοναδική μεταβατική περίοδο. Δεν θέλετε να αλλάξει η κατάσταση πολλέ φορέ. Και ξέρω ότι πολλοί ακούν αυτήν την ε, συνεδρίαση της Επιτροπής μας σήμερα από το Λονδίνο και από τις Βρεξέλλες. Είναι σημαντικό λοιπόν το στοιχείο αυτό της μίας και μοναδικής αλλαγής. Μία ερώτηση. Στη Μεγάλη Βρετανία παράγονται αυτοκίνητα Toyota. Τα αυτοκίνητα αυτά πριν ε, περάσουν στην εξαγωγή, περνούν από εσά. Και τι θα σημαίνει αυτό στο μέλλον σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα εισαγωγής και απαντήστε αν θέλετε. Όχι, δεν είναι δύσκολο Όντως υπάρχουν αυτοκίνητα διάλευσης ε, πάρα πολύ σημαντικά που έρχονται σε εμά, ε, στο, περνάνε στον Εμένο Βασίλειο για να ε, πάνε μετά στη Χιλή και αλλού. Και έχουμε και αυτοκίνητα από την Ιαπωνία για το Ηνωμένο Βασίλειο που περνούν από το λιμένα μας. Έχουμε μεγάλο όγκο. Το τελευταίο που είπα είναι ότι έχουμε ένα εκατομμύριο αμάξια που συνδέονται με το Ηνωμένο Βασίλειο και 150.000 που είναι διεθνές εμπορεύματα, διεθνή εμπορεύματα και περνούν από το λιμένα. Είναι σημαντικό να κρατήσουμε αυτή την προστιθέμενη αξία στην φάση μετά το Brexit. Δεν είναι δύσκολο, αλλά προφανώς εξαρτάται από τις πολλές συμφωνίες που θα πρέπει να κάνουμε με τα Τελωνία. Πώς θα κατηγοροποιούνται τα αυτοκίνητα αν πλένονται, αν ε, αλλάζει κάτι, αν ε, ε, ενισχύονται κτλ. Μάλιστα, μία ερώτηση προς τον κύριο Λάιτον. Οι Βρετανικοί λιμένε νόμιζαν ότι είναι ιδιωτικοί, ότι δεν είναι κρατική ιδιοκτησία, δεν είναι δημόσια ιδρύματα, είσαστε απλέ επιχειρήσει. Αυτό σα δίνει πιο πολύ περιθώριο για να συνεργαστείτε με το Δουβλίνο σε σχέση, για παράδειγμα, με ένα δημόσιο λιμάνι όπως είναι το Ζεμπρίχε ή το Ρότερνταμ. Απάντηση. Ναι, κοιτάξτε. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται περιθώριο, περιθώριο δράσης. Αλλά ναι, είναι ιδιωτικοί οι πιο πολλοί λιμένες. Υπάρχουν και κάποια δημόσια λιμάνια όμως. Το Ντόβερ είναι ένα δημόσιο λιμάνι. Περιθώριο δράσης λίγο πολύ αυτά που είπε ο συνάδελφος σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την επαφή με τις ε, Βρετανικές αρχές. Νομίζω ότι όλοι είναι σε στενό διάλογο με την Βρετανική κυβέρνηση, είτε είναι ιδιωτική είτε δημόσιοι λιμένες. Ε, μία ερώτηση προς την κύριο O'Reilly. Μέσα του Δουβλίνου έρχονται προϊόντα που πάνε στο λιμένα του Μπέλφας. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Πολύ απλά δεν ξέρω. Είναι ένα από τα μεγάλα ερωτηματικά της πρώτης φάσης. Πολύ καλή ερώτηση το θέμα των χερσαίων συνόρων και το θέμα της Ιρλανδίας. Είναι ένα πραγματικά ε, πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Δεν εμπιπτεί καθόλου στον τομέα των αρμοδιοτήτων μου. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Στην παρούσα φάση πολλά αγαθά από το λιμάνι του Δουβλίνου και έρχονται από το, τη Βόρεια Ιρλανδίνα γιατί πολύ απλά έρχονται από τον Ατοταπλία, πάνε βόρεια στην Ιρλανδική θάλασσα και είναι λίγα τα χιλιόμετρα μεταξύ Belfast και σε πολλές ε, και Δουβλίνου. Και δεν ξέρω πραγματικά τι θα γίνει. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε στο λιμάνι του Δουβλίνου είναι να δημιουργήσουμε τις υποδομές. Πιο πολλά δεν μπορούμε να κάνουμε και ελπίζουμε να παραμείνει ανοιχτό το σύνορο αυτό για όλους και για τα αγαθά και για τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Φανεκόμπ ή κυρία Άντερσον. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ράιλι, πολύ χάρηκα που άκουσα την εισήγησή σας, όλων σας και ε, σύντομα θα επισκεφτούμε το Δουβλίνο ε, με προσωπία της Τραν πολύ σύντομα. Χαίρομαι πολύ που είσαστε τόσο αισιόδοξε, αλλά εγώ έχω σημαντικές αμφιβολίε αν είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα για λιμάνια του Ηνωμένου Βασιλείου. Όσον αφορά όμως την νομοθετική ρύθμιση, ο κανονισμός ε, που συζητήσαμε εδώ στην Επιτροπή μας, ε, πιθανότατα να γνωρίσετε ότι ήταν πολύ επίμαχο ζήτημα εδώ στο Κοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά καταλήξαμε σε πολύ καλό και ισορροπημένο αποτέλεσμα με μέτρα σχετικά με την διαφάνεια, ε, τι επενδύσει και την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού. Τα βρετανικά λιμάνια λένε τώρα στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ότι δεν θέλουμε να εφαρμόσουμε τον κανονισμό αυτόν και έτσι δεν θα υπάρχουν συνθήκες ανταγωνισμού. Πώς το βλέπετε αυτό? εκτιμώ πολύ ε, τους λιμένες ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, είναι, λιμάν, είναι νησί με πάρα πολλά λιμάνια, λειτουργεί πολύ καλά. Εμείς όμως χρησιμοποιούμε διαφορετικό πρότυπο στην Ιρλανδία και νομίζω ότι αυτή είναι η φύση και γενικά των λιμένων ε, υπάρχουν διαφορετικές δομές σε διάφορα μέρη. Εγώ δεν ε, ανησυχώ ότι ε, το διαφορετικό ρυθμιστικό πλαίσιο για το Ηνωμένο Βασίλειο θα επηρεάσει τους λιμένες της Ιρλανδίας. Η μόνη περίπτωση είναι αυτό που ανέφερα νωρίτερα. Ναι, συμφωνώ ότι πιο σημαντικό για μας ε, είναι, ο εκτελονισμός, οι τελωνιακές διασαφήσεις και είναι πολύ σημαντικό να λειτουργήσει ακριβώς αυτό το σύστημα, να δούμε τι θα πρέπει να δηλώνεται, πόσες φορές αν ε, μεταφέρεται πέρα δόθε και να έχουμε συνθήκες ίσου ανταγωνισμού. Και θα ήθελα να προσθέσω αυτό που είπε και ο κύριος Φαντεκάμπ, που επίσης ε, σημαντικό δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικά καθεστώτα στις κάτω χώρες, ε, το Βέλγιο και την Ιρλανδία για παράδειγμα. Ε, η κυρία Άντερσον, ε, κύριε Λέιτον, ε, φαίνεστε πολύ αισιόδοξο ότι θα υπάρξει ρυθμιστική ευθυγράμμιση και γι' αυτό ε, δεν ε, θα είναι η τελωνιακή έλεγχη πρόβλημα. Μήπως όμως ε, μπορείτε να σχολιάσετε το γεγονός ότι θα είμαστε πια τρίτη χώρα όσον αφορά την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι τόσο χαλαρή όσον αφορά την ε, διαφορετική ε, διενέργεια των ε, τελωνιακών ελέγχων. Τα αγαθά που θα έρχονται μέσω Ηνωμένου Βασιλείου, που θα είμαστε πια τρίτη χώρα, θα υπόκεινται σε διαφορετικά πρότυπα. Εάν υπάρξει, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα υπάρξει ρυθμιστική ευθυγράμμιση, αλλά όπως και να έχει, πώς το βλέπετε ε, κάποιες παρατηρήσεις ήδη από την πρώτη μέρα εάν δεν υπάρχει ρυθμιστική ευθυγράμμιση αυτά που κάνουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την υγεία φυτών, ε, τα κτηνιατρικά θέματα κτλ θα συνεχίσουν να ισχύουν όπως και πριν το Brexit. Δεν ε, θα πρέπει να υπάρξει ανησυχία λοιπόν για τέτοιου είδους ελέγχους. Σε πολλά χρόνια από τώρα, αν υπάρξει απόκληση των προτύπων και εφαρμόσουμε ε, απαιτήσει ανάλογα με το τι εμπορικές συμφωνίες θα έχουμε τότε ε, σημαίνει παρόλα αυτά ότι θα υπάρχει αρκετός χρόνος ε, προσαρμογής ε, και οι παρατηρήσει μου επικεντρώνονται πιο πολύ στην, στο, στο εγγύς μέλλον. Το μόνο που θα μπορούσα να προσθέσω είναι ότι είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε αυτό που είπα νωρίτερα. Με το καθεστώ που έχουμε αυτή τη στιγμή, με απόκληση των διαφόρων προτύπων στα διάφορα μέρη του κόσμου, χάρη στα συστήματα τελωνιακή διασάφηση που έχουμε αυτή τη στιγμή, οι αρχέ του Ηνωμένου Βασιλείου σταματάνε μόλις το 1,3% των αγαθών που εισέρχονται στη χώρα. Ε, αν ε, αφαιρέσετε ακόμα και το 80 ή 40% αυτού του ποσοστού, δεν μπορώ να φανταστώ κάποια σωστή ρεαλιστική προσέγγιση που να οδηγήσει σε σταμάτημα, σε μπλοκάρισμα των διαδικασιών. Όσον αφορά το ντόβερ, θα πρέπει να μειώσουμε τον χρόνο των ελέγχων σε 15 δευτερόλεπτα για να αποφύγουμε ε, τη συμφόρηση, τις ουρές και το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει ότι μπορεί να εφαρμόσει τεχνολογίες που να μειώσουν το χρόνο στα δύο λεπτά, αλλά αυτό δεν αρκεί καθόλου για τον Dover. Πώς θα γεφυρώσουμε λοιπόν το χάσμα ανάμεσα στα δύο λεπτά και τα 15 δευτερόλεπτα. Ναι, έχετε δίκιο και η ABP ε, διαχειρίζεται το λιμάνι του Ντόβερ και καλύτερο να απαντήσει μόνη της, αλλά το λιμάνι του Ντόβερ. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεργαστεί στενά με την κυβέρνηση και θα καταλήξει σε κάποια λύση. Δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή η λύση, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται και θα φροντίσει να υπάρχει κατάλληλο σύστημα. Επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι εδώ. Δεν νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν επιπλέον έλεγχοι. Μπορεί να λέτε ότι δεν είναι απαραίτητοι, αλλά θα υπάρξουν. Όταν κάποιο βρίσκεται εκτό τη Τελωνιακή Ένωση, θα πρέπει να έχει κάποιο σύστημα για ελέγχου. Θα χρειαστεί λοιπόν κατάρτιση του προσωπικού. Ε, αυτή τη στιγμή έχουμε πέντε ανθρώπου που σπουδάζουν εκτελονισμό, αλλά θα χρειαστούμε εκατοντάδε για να στηρίξουν ένα τέτοιο σύστημα. Ίσως ε, λοιπόν είναι σημαντικό να γίνουν επενδύσεις ε, και στην κατάρτιση ανθρώπων που θα μπορέσουν να δημιουργήσουν ε, συστήματα λειτουργικά και μία διευκρίνηση. Δεν είπα ότι δεν θα χρειαστούμε καθόλου επιπλέον ελέγχους, απλά επισημαίνω ότι οι επιπλέον έλεγχοι που θα χρειαστούν δεν θα οδηγήσουν σε συμφόρηση του συστήματος. Αυτό προσπαθώ να πω. Ευχαριστώ. Κυρία Μάισνερ, για πέντε λεπτά. Και συνέχεια κυρία Ζουλεμβάνης. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση προς τον κύριο Κούντς και προς τον κύριο Λέιτον κυρίως. Ήδη βλέπουμε αλλαγή στην οικονομία. 50% του διεθνού εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 40% περνάει από τα λιμάνια. Αν υπάρχει λιγότερη παραγωγή στην Ηνωμένο Βασίλειο, σε ό,τι αφορά την ε, ε, γερμανική παραγωγή της Siemens, για παράδειγμα. Αυτά δεν εξαγάγονται εκ νέου και δεν θα μπορούσαν τελικά επιπλέον έλεγχοι εισαγωγών και εξαγωγών να οδηγήσουν στην ύπαρξη λιγότερων επιχειρήσεων. Αυτό δεν σας απασχολεί σε ό,τι αφορά και τους ε, Βρετανικούς λιμένες. Ευχαριστώ να απαντήσω εγώ πρώτα. Όχι, δεν φοβόμαστε. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο κουραστικές οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σε κάποιες περιπτώσεις. Είτε ανησυχούμε είτε όχι. Σε τελική ανάλυση το αποτέλεσμα των μερωτικών εμπορικών διαπραγματεύσεων είναι αυτό που θα μετρήσει και αυτές οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μπορεί να λάβουν χώρα σε πνεύμα καλής θέληση προκειμένου να υπάρξει κοινή ευημερία, αλλά ενδεχομένω να λάβουν χώρα και σε διαφορετικό πλαίσιο δεδομένης όμως της στενής συνεργασίας με τους συναδέλφου ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και δεδομένης και της συνεργασίας με τη Siemens που είναι ένας από τους μεγαλύτερου ε, πελάτες δεν έχω που ανησυχίε. Ναι, κοιτάξτε και από πλευρά μα. Ε, φόβος, ο φόβος δεν είναι καλός σύμβουλος ε, και καλός, ε, καλό είναι πάντα πιστεύω να υπάρχουν καλές σχέσεις με τους γειτονικέ χώρες και αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι δεν θα υπάρξουν αναταραχές βραχυπρόθεσμα σε κάποιους οικονομικούς κλάδους. Αυτό φυσικά εξαρτάται και από άλλους ε, φορείς, για παράδειγμα, στο τιμία μεταξύ ε, λίρας και ευρώ. Ο τομέας της φαντουργίας των τροφίμων, όπως είπατε, πολύ ευαίσθητος. Νομίζω όμως ότι σε βάθος χρόνου η κατάσταση θα διαμορφωθεί όπως είναι διαμορφωθεί. Σας ευχαριστώ να απαντήσω, στα, να κάνω την ερώτηση στα αγγλικά προς τον κύριο Λέιτον σε ό,τι αφορά τα βρετανικά λιμάνια. Πιστεύετε ότι υπάρχει πλεονέκτημα από το Brexit, δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οποιασδήποτε κανονισμοί για τη παροχή υπηρεσιών στους λιμένες ή, εν πάση περιπτώσει, δεν θα περιορίζεται και από άλλους κανονισμούς. Θα είσαστε πιο ελεύθεροι και μήπως είναι μειονέκτημα να μην συμμετέχετε στους διαδρόμους τι και τι υπερισχύει από τα πλανεκτήματα ή τα μειονεκτήματα. Um, I really... Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει συζήτηση με εικασίε για τα ενδεχόμενα πλανεκτήματα και μειονεκτήματα βάσει διαπραγματεύσεων που δεν ξέρουμε πώς διαμορφώνονται στην παρούσα φάση, πόσο μάλλον το αποτέλεσμά του και η έκβασή του μπορώ να σας πω 20 ενδεχόμενα πλεονεκτήματα και 20 καζόμενα μη μειονεκτήματα. Όλα αυτά αποτυπώνουν τις πολιτικές μας απόψεις ενδεχομένως, αλλά με πάσα ειλικρινία δεν έχω έρθει εδώ να κάνω αυτό. Εγώ έχω έρθει να μιλήσω, για την ενδεχόμενη αντίκτυπο στη ροή των εμπορευμάτων. Μάλιστα, μία ερώτηση προς τον κύριο Ρέιλι. Έχω μιλήσει με διάφορου εκπροσώπου στον τομέα των μεταφορών στην Ιρλανδία που φοβούνται ότι μπορεί να υπάρξει μεγάλο αντίκτυπο στην Ιρλανδία από τον Brexit, να επηρεαστεί το εμπόριο μεταξύ τη Ιρλανδία και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά φαίνεται ότι εσεί δεν φοβάστε το ίδιο για τα λιμάνια ή πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να πλήξει και του λιμένες. Αν κατάλαβα σωστά, δεν θεωρείτε ότι θα υπάρξουν προβλήματα. Ευχαριστώ για την ερώτησή σα, γιατί θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι πολύ σημαντικό όταν μιλάω για το ότι δεν φοβάμαι τον αντίκτυπο του Brexit. Μιλάω αποκλειστικά και μόνο για το λιμάνι του Δουβλίνου. Θα υπάρχουν. Το πρώτο που θα πω για το Brexit είναι ότι δεν θα έχει ως αποτέλεσμα πιο πολύ εμπόριο. Θα υπάρχουν τμήματα της Ιρλανδικής οικονομίας που θα πληχθούν ιδιαίτερως ε, Έχουμε μια μεγάλη βιομηχανία, για παράδειγμα, που περνάει από τους λιμένες το μέσο των τροφίμων της Γεωργίας σίγουρα θα πληχθεί. Μπορεί να ανακάμψει σε βάθος χρόνου, αλλά σίγουρα για μία περίοδο θα υπάρξουν απώλειες θέσεων εργασίας και αρνητικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις και δεδομένες και του τομέα εφαρμογής ε, της ε, Επιτροπής σας. Θα κοιτούσα και το δομέα της μεταφοράς φορτίων στην Ιρλανδία. Ως τώρα είμαστε γύρω στις 20 ώρες για τη μεταφορά φορτίων. Αυτό στο μέλλον φαντάζομαι δεν θα ισχύει στο μέλλον. Και έτσι θα πρέπει να ξεκινήσουν άλλες διαδικασίες λες και περνάει κανείς μέσω Κίνας, μέσω Αφρικής. Αυτή θα είναι η πραγματικότητα των ελέγχων. Θα είναι λοιπόν πολύ σημαντικές αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις ε, για την Ιρλανδική οικονομία. Για το λιμένα του Δουβλίνου νομίζω ότι δεν θα υπάρξει ιδιαίτερος αντίκτυπος, ε, γιατί πολύ απλά έχουμε άλλες ανάγκες, όπως την αντιφορτική κατάστασή μας στην κρίση του 2018 η κυρία Ζιλ Εβέντς για πέντε λεπτά και μετά ο κύριος Καν. Um, Ευχαριστώ πολύ. Εκπροσωπώ την Ουαλία και φυσικά θα υπάρχει μεγάλος ε, αντίκτυπος, ιδιαίτερα στο λιμένα Holyhead, που έχει τα μεγαλύτερα φέρη της Ευρώπης αυτή τη στιγμή και δεν έχει την δυνατότητα και τη χωρητικότητα ε, τη δυνατότητα περισσότερο σε αυτή την περίπτωση να κάνει όλους τους ελέγχους αν αποτελέσει σκληρό σύνορο. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσουμε τις καλές μας σχέσεις με την Ιρλανδία. Έχει γίνει μια έρευνα από την τοπική κυβέρνηση για το μέλλον αυτού του λιμανιού και αυτό που ε, μας ενδιαφέρουν είναι τα ελεύθερα λιμάνια, οι ελεύθερες ζώνες που προτάθηκαν για να αντισταθμίσουν τις ε, αρνητικές συνέπειες μιας, ενός σκληρού Brexit. Θα ήθελα τα σχόλιά σας. Το Holyhead είναι ένα λιμάνι που θα αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα με το Dover. Ε, ήθελα όμως να τονίσω ότι βράχει πρόθεσμα μπορούμε να αντιπαρέλθουμε τα προβλήματα. Ε, έχει σημασία η προσέγγιση των κυβερνήσεων και από τις δύο πλευρές. Ε, εάν σταματάμε κάθε φορτηγό, γιατί αυτή είναι η προσέγγιση, τότε είναι πρόβλημα. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ που θίξε το θέμα των ελευθέρων εμπορικών ζωνών. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει σε πολλούς κύκλους για μετά το Brexit είναι κάτι που ίσως θα δημιουργήσει την αναδιάρθρωση και τον ανασχηματισμό των ε, λιμένων. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις βιομηχανικές δραστηριότητες και τις, ε, την κατασκευαστική, τον κατασκευαστικό τομέα. Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε βεβαίως και να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Το λιμάνι του Holyhead είναι παρόμοιο με του Δουβλίνου, όπως ισχύει στη σχέση Dover-Καλέ. Αυτό είπαν ε, και στην Ιρλανδία ως προς την τελωνιακή σχέση. Εάν ε, γίνουν τελωνιακοί έλεγχοι με την παρούσα ε, τάση που διαγράφεται θα είναι πολύ περιορισμένοι. Θα πρέπει να υπάρχουν ε, διοικητικά έξοδα, γενικά έξοδα, τα οποία θα ξαναμπούν ενώ είχαν βγει μετά το 1992. Είναι ε, μία πραγματική πρόκληση ιδιαίτερα για τον διάπλου μεταξύ Δουβλίνου και Χόλιχετ που διαρκεί 3,5 ώρες γιατί ε, νομίζω ότι οι συγκεκριμένες ε, αλυσίδες προμήθειας, εφοδιαστικές δηλαδή, θα πρέπει να περάσουν από το ε, Holyhead στο Σέμπρουχε ή στο Ρότερνταμ. Άρα ίσως αυτή η εφοδιαστική πορεία να αλλάξει. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι γίνεται στο Δουβλίνο ας πούμε με αγαθά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να ισχύσουν επί πέντε λόγω του μεγάλου φόρτου. Ο Ντέιβιτ μίλησε για 1,5%. Αν έχουμε δύο ελεύσεις από το Holyhead, θα έχουμε να κάνουμε με μία αύξηση εις πενταπλούν. Ε, θα μπορούσαμε να έχουμε δηλαδή 50 φορτία τα οποία θα πρέπει να ελεγχθούν. Δείτε λοιπόν πώς θα γίνει αυτός ο κατακερματισμός. πολλές φορές ε, ξεφεύγουμε γιατί μας ενδιαφέρει βεβαίως, ε, μας ενδιαφέρουν οι συνταρακτικοί τίτλοι ή τα πολιτικά σενάρια. Αλλά νομίζω ότι το σενάριο μετά το Brexit δεν είναι τόσο αρνητικό για τους λιμένες. Ως προς τις ελεύθερες ζώνες μεταφορών με τελωνιακές υπηρεσίες υπάρχουν δύο στοιχεία αν τα αγαθά προέρχονται από, το, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή εκτός και μεταβαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν προέρχονται εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταβαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, τότε θα πρέπει να έχουμε μια ελεύθερη ζώνη όπου αναστέλλεται η τελωνιακή δήλωση. Αυτό ήδη συμβαίνει τώρα, αλλά τώρα υπάρχει τελωνιακή ένωση για τα αγαθά από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν δύο στοιχεία. Καταρχήν να υπάρχει η τελωνιακή δήλωση από τις χώρες εξαγωγής για τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά για τις μικρότερες θα υπάρχει μεγαλύτερος φόρτος Γι' αυτό θα πρέπει οι ζώνες να αφορούν τους λιμένες και από εκεί να οργανώνονται οι εξαγωγές. Διαφορετικά θα εξαφανιστούν πολλές μικρές επιχειρήσεις γιατί δεν θα μπορέσουν πια να διαχειριστούν αυτές τις μεταφορές. Οι μεγάλες θα τα καταφέρουν, αλλά για τις μικρότερες θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ζώνη στο λιμένα για τις δηλώσεις εξαγωγών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε υπερβεί το χρόνο, το χρόνο μας. Ο κύριος Κάντς έχει το λόγο για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν χρειάζομαι τρία λεπτά. Θα είμαι πιο σύντομος. Πολύ σύντομε ερωτήσεις έχω. Σας ευχαριστώ που μας δώσατε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη σημερινή ακρόαση. Η ερώτησή μου απευθύνεται στον κύριο Λέιτον. Οι εφοπλιστές ε, τη της Βρετανίας ε, φοβούνται ότι θα χάσουν ε, μέρος του εμπορίου με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα ήθελα λοιπόν σε συνέχεια αυτών που είπαν οι συνάδελφοι να ρωτήσω τι όφελος θα έχει το Ηνωμένο Βασίλειο με την αποχώρηση του από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά ε, το εμπόριο και προβλέπεται ε, ναυτιλιακές γραμμές να αποφεύγουν τους λιμένες του Ηνωμένου Βασιλείου. Νομίζω ότι γενικά είμαι ενδιαφέρον άνθρωπο ε, στι συζητήσει μου, αλλά σήμερα μάλλον επαναλαμβάνομαι. Δεν μπορώ να απαντήσω σε τέτοιε ερωτήσει. Μπορούμε να κάνουμε υποθέσει. Αλλά απομένουν πολλά να διευκρινιστούν. Ε, έχουμε πολλά να μάθουμε ακόμα όσον αφορά την πορεία των διαπραγματεύσεων που όπως είπα μπορεί να διεξαχθούν σε επικοδομητικό κλίμα ή όχι. Ίσως λοιπόν θα είναι πιο χρήσιμο να το ρωτήσετε αυτό ε, στο μέλλον. Ε, ζητώ συγγνώμη για την απάντησή μου, ελπίζω λίγο να σας βοήθησε. Να επανέλθω σε αυτό κύριε Λέιτον. 57 εβδομάδες απομένουν. Ναι, ακούμε συχνά στο, στις ειδήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι το ρολόι τρέχει. Αλλά τι, να πω, πρέπει να είναι πάρα πολύ ενοχλητικό αυτό το ρολόι για τον κύριο Μπαρνιέ. Η κυρία Κλούν, έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λέιτον. Ήθελα και εγώ να αναφερθώ στο ρολόι και τους λιγότερο από 13 μήνες που απομένουν. Ακούσαμε ε, τον Λιμπένα του Ρότερνταμ να προετοιμάζεται για, ε, για το χειρότερο ενδεχόμενα. Ο, ο Μάρτιος του 2019 πλησιάζει και προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο το Ηνωμένο Βασίλειο να βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα πρέπει να κλείσει κάποιες ε, υπηρερίες. Μας μιλήσατε για ποσοστά 55%, 45% στη χειρότερη περίπτωση τον Μάρτιο του 2019 το 100% του εμπορίου σας ε, θα ε, προέρχεται από εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είσαστε αισιόδοξο, ε, πιστεύετε ότι η ρυθμιστική ευθυγράμμιση θα ισχύσει από την πρώτη μέρα, αλλά... Εγώ ως Ιρλανδί σκέφτομαι τους μεταφορείς, τους διάφορους φορείς εάν δεν υπάρχουν ε, οι υποδομές για το χειρότερο ενδεχόμενο για τον Μάρτιο του 2019. Τι θα γίνει, διότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου λέει ότι θέλει να βρίσκεται εκτός της εσωτερικής αγοράς και εκτός της Τελωνιακής Ένωσης. Φαίνεται να είστε πιο αισιόδοξος και είπατε ότι θέλετε καλές σχέσεις με τους άλλους ευρωπαϊκούς λιμένες, τους γειτόνους σας. Αλλά και οι λιμένες αυτοί θα πρέπει να προσαρμοστούν, να προσαρμόσουν τις ε, υποδομές τους άσχετα από το τι φιλικές σχέσεις διατηρείτε. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας αυτή. να κάνω μία πολύ απλή σύγκριση. Έχουμε αρνίσιο παϊδάκι. Και την ημέρα πριν το Brexit, το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την επόμενη μέρα ε, αυτό δεν θα αλλάξει. Θα συνεχίσει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσει. Εάν λοιπόν είμαστε ρεαλιστές και αν ε, ακολουθήσουμε μια προσέγγιση που να βασίζεται στον κίνδυνο, ε, δεν θα κλείσουμε τα πάντα και μπορεί ναι, να είμαι αισιόδοξο στο θέμα αυτό. Νομίζω όμως ότι ιδιαίτερα σαφές σήμερα το απόγευμα ήταν ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές ώστε να διατηρηθεί το εμπόριο προς όφελος της οικονομίας και αυτό τελικά θα πρέπει να μας κάνει αισιόδοξου. Έτσι μπορεί να συνεχιστεί το εμπόριο και να έχουμε ανάπτυξη. Μπορεί φυσικά να βλέπει τα πράγματα κανείς από διαφορετική οπτική, αλλά δεδομένων των κοινών οικονομικών συμφερόντων που έχουμε, θα πρέπει όλοι να επιδιώξουμε μια λογική λύση. Και το θέμα δεν είναι αν είναι κανείς αισιόδοξο ή απεσιόδοξος. Αλλά το ότι κάποιο βρίσκεται εκτό τη Θελωνιακή Ένωση δεν σημαίνει ότι θα, γίνεται, θα επικρατεί χάο στα σύνορα. Εάν δούμε κάτι τέτοιο, αυτό θα είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα πολιτικών ε, αποφάσεων. Εγώ αυτό που ακούω είναι ότι εύχεστε, ελπίζετε, αλλά δεν σχεδιάζετε για πανενδεχόμενο. Ναι, να συμπληρώσω. Αυτό που ακούει κανεί από συναδέλφου σε όλου του τομεί είναι ότι υπάρχει μια σειρά σεναρίων. Χρήσιμο είναι να προετοιμαστεί κανεί για όλα αυτά τα ε, ενδεχόμενα και νομίζω ότι ο κύριος από το Ρότερδαμ ε, ήταν πολύ εύστοχος. Μου ζητήσατε να σχολιάσω σχετικά με την αισιοδοξία για απεσιοδοξία, αλλά νομίζω ότι όλα τα γεγονότα μας οδηγούν στην αισιοδοξία. Ε, Έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Ο κύριος Πέιλι. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επανέλθω στα τελωνιακά. Πολλά προελέχθησαν αλλά ο κύριος ε, ο Ράιλι μίλησε για νέα βιομηχανία διοικητικών εξόδων το οποίο σημαίνει μεγάλη κατασπατάληση χρημάτων. Έχετε λοιπόν αρνητική άποψη για τις καθυστερήσεις και θα πρέπει να, μας το, να το δούμε σε 57 εβδομάδες. Ο κύριος ε, Κούνς ε, μίλησε για την ψηφιακή πλατφόρμα η οποία θα μπορέσει να λύσει πολλές από αυτές τις διατυπώσεις για να αποφύγουμε αυτές τις καθυστερήσεις και τις σχετικές ζημιές. Άρα πού βρισκόμαστε, ε, μιλάμε για την ψηφιοποίηση όλων αυτών των διατυπώσεων. Αυτό θα μπορούσε να αποσοβήσει τους κινδύνους. Βεβαίως, η τεχνολογία και οι ψηφιακές διαδικασίες θα καταστήσουν φθηνότερα, χαμηλότερα τα γενικά έξοδα. Ο Πάλο Τσετσίνη το 1991 ο Ιταλός αυτός οικονομολόγος ε, μίλησε για μεγάλο κέρδος από την άρση αυτών των ελέγχων εμείς τώρα θεωρούμε ότι θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τα ε, γενικά έξοδα και το χρόνο με τις νέες τεχνολογίες. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα παϊδάκια της Δευτέρας είναι τα ίδια με τις Τρίτης, αλλά υπάρχουν νέες προαπαιτήσεις πριν μπουν στο πλοίο και σταλούν αλλού. Και γι' αυτό μιλάμε για προετοιμασίες στο Δουβλίνο. Αυτό αφορά τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατέστησαν λειτουργική και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να προσθέσω ότι εάν συγκρίνουμε την κατάσταση με το Ρότερταμ, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι μας έχει καλομάθει η Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό δεν υπάρχει ψηφιοποίηση. Θα πρέπει να επιταχύνουμε το, τα συστήματα όπως ισχύουν στην ανοιχτή θάλασσα. Έτσι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι εύκολη η θέση εφαρμογή εγκαίρως. Η κυρία Φώστερ, για τρία λεπτά. Θα είμαι πολύ σύντομη. Λυπάμαι που δεν, είμαστε, που δεν ήμουνα σε όλες σας τις παρουσιάσεις. Εγώ θεωρώ ότι το ποτήρι είναι μισογεμάτο ε, λήφθη μια απόφαση δημοκρατικά και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες. Ε, είμαι από τους πολιτικούς που πιστεύουν ότι πάντα υπάρχει μία απάντηση. Διαφορετικά δεν θα πρέπει να είχαμε διαλέξει την πολιτική. Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι θέμα και πολιτικής θέλησης. Βεβαίως υπάρχουν προκλήσεις, αλλά νομίζω ότι αυτό που δεν αναφέρθηκε είναι ε, η εργασία στα λιμάνια, ε, στη βιομηχανία, ε, από τις θαλάσσιες μεταφορές. Υπάρχουν λοιπόν όλοι οι οργανισμοί που θα πρέπει να διευκολύνουν την μετάβαση για το Brexit το Μάρτιο του χρόνου. Νομίζω ότι ε, υπάρχει, υπάρχουν οι εγκέφαλοι και εδώ και αλλού έτσι ώστε να λύσουμε τα ζητήματα. Δεν πρέπει λοιπόν να είμαστε αισιόδοξοι παρά τις ε, προκλήσεις διαφορετικά. Δεν θα κάνουμε παρά μία τρύπα στο νερό και κανένας δεν θα θέλει να έρθει ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Ιρλανδία για να βρει λύσεις. ξέρω ότι θα πρέπει να εξευρεθούν λύσεις γιατί εμείς έχουμε ένα από τα πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά λιμάνια στον κόσμο όπως ε, γνωρίζετε όλοι. Να είμαι πεπισμένος ότι θα τα καταφέρουμε γιατί είχαμε ιστορικές εμπορικές σχέσεις και θα συνεχίσουμε. Τώρα το ζήτημα είναι της αφήνειας Ποιος είναι ο πιο διαφανής τρόπος λειτουργίας. Υπάρχει απόφαση, αλλά υπάρχει ασάφεια ε, αν θα υπάρχει εμπορική συμφωνία, πώς θα έχουν τα τεχνικά ζητήματα τελωνιακών ελέγχων και ούτω καθεξής. Γι' αυτό θα πρέπει να ορίσουμε τη μεταβατική περίοδο, γιατί δεν θα είμαστε έτοιμη μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους. Από τη φύση μας είμαστε αισιόδοξοι σήμερα, λέμε ότι υπάρχουν πραγματικότητες που μας απασχολούν. Είναι δύσκολο για τους ε, ανθρώπους ε, επιτόπου, που εργάζονται επιτόπου να βρουν ε, λύσεις. Γι' αυτό θα πρέπει σε αυτή τη φάση να προετοιμαστούμε δηλαδή να προετοιμαστούμε για το χειρότερο και να περιμένουμε το, και να ελπίζουμε για το καλύτερο για το μόνο που είμαι σίγουρος είναι ότι δεν θα υπάρξει αξίση εμπορίου. Δεν θα ζήσουμε τον κατακλυσμό του 2008, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε αρνητικές απόρριες, περισσότερα έμεσα έξοδα, αλλά φυσικά το ποτήρι είναι μισογεμάτο και θα τα καταφέρουμε στα λιμάνια μας. θα έχετε παρατηρήσει και αναφέρθηκα στα παϊδάκια για ένα συγκεκριμένο λόγο. Θα έχετε λοιπόν παρατηρήσει ότι είναι θέμα πολιτικής θέλησης και κινήτρων κατά τις διαπραγματεύσεις φυσικά από τεχνικής πλευράς το εμπόριο θα ρέει και θα αναπτύσσεται. Το ζήτημα είναι ποιοι είναι οι στόχοι αυτών που προωθούν τις διαπραγματεύσεις και είναι επικεφαλής. Ε, κυρίες, ολοκληρώνεται αυτή η συνεδρία, η ακρόαση. Να ευχαριστήσω τους τρεις προσκεκλημένους μας για την ποιότητα της συζήτησης και δεν θα πάρω το παράδειγμα με το παϊδάκι. Θέλω να τρώω λιγότερο κρέα. Το θέμα δεν είναι αν είμαστε αισιοδοξοί ή απεσιοδοξοί. Το θέμα είναι να είμαστε ρεαλιστέ. Tout le monde peut être euh, dans un... Voilà, on peut être optimiste de... Γιατί η αισιοδοξία και μόνη της δεν αρκεί. Δεν θα λύσει τίποτα. Δεν θα μας βοηθήσει ενώπιον των προκλήσεων. Έχουμε ακούσει συναδέλφου και από τον τομέα των αερομεταφορών και από τον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών και τώρα και εσά. Όλο ο κόσμο ανησυχεί. Τι θα συμβεί. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο συμφωνήσαμε όλοι σήμερα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ε, μεταβατική περίοδος. Αλλά μία φορά. Και εδώ Συμφωνούμε να μην αλλάζουμε κάθε έξι μήνες για να καθοριστεί ο οδικός χάρτης. Και επίσης συμφωνούμε και για άλλα στοιχεία. Αν υπάρχουν έλεγχοι, για παράδειγμα, θα πρέπει να απλοποιήσουμε τα, το διοικητικό σκέλος. Δεν το συζητήσαμε αυτό επιθαμένως. Θυμάμαι όμως ε, για τις ανησυχίες που εκφράστηκαν σε ό,τι αφορά την αύξηση του διοικητικού άκτους. Εσείς από τους λιμένες θα πρέπει να απαλύνετε αυτό το άχθος. Γιατί ενδεχομένω να χρειαστεί να καλυφθούν αυτές οι τεράστιες ε, ουρές που θα σχηματιστούν. Αυτά είναι λοιπόν κάποια ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να λάβουν απαντήσεις κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο. Σε αυτή τη, με αυτή την αχτίδα, αν θέλετε, ρεαλισμού. Ελπίζουμε να έχουμε μια κοινή πλατφόρμα για τις κοινέ αξιώσεις, να τα θέσουμε όλα αυτά επιτάπητος για να μην μας πιάσει εξαπίνης ο Μάρτιος του 2019. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή μου. Θα σας χαρούμε να σας ξαναδούμε σύντομα. Είστε ευπρόσδεκτοι. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν που μας θυμήσατε με την εμπειρογνωμοσύνη σας αλλά και με το χρόνο σας. écoutez, vous avez aimé le secteur maritime, vous allez adorer. Αν ναι, σα άρεσε η προηγούμενη συζήτηση, θα λατρέψω την επόμενη. Για τον τομέα των αερομεταφορών. Καλώ ήλθατε, κύριε Κορνελή. Allez, Allez, nous continuons. Να συνεχίσουμε με την έκθεση του κυρίου Πίπερ για τη του ανταγωνισμού στον τομέα των αερομεταφορών. 288 οι τροπολογίε που κατέστηκαν. Θα δώσω φυσικά το ρόλο στον εισηγητή μας και μετά θα ακολουθήσουν οι σκιώδεις εισηγητές και όποιο άλλο θέλει να πάρει το λόγο στο τέλος, θα δώσω το λόγο προφανώς και στον κύριο Κορνέλη ο οποίος είναι εδώ. Για να μας δώσει την άποψή του για την έκταση. Κύριε Πίπερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα διαρκέσει πολύ η εισήγησή μου. Έχουμε κοιτάξει τις τροπολογίες, όπως είπατε, περίπου 300 είναι στον αριθμό. Δεν είναι φρικτός ο αριθμός. Και υπάρχουν ε, και τροπολογίες που είναι πολύ παρόμοιες προς το περιεχόμενο. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιες είναι πολύ αμφιλεγόμενες. Άρα, διαπιστώνουμε ότι στο Κοινοβούλιο χρειαζόμαστε ένα ισορροπημένο κείμενο, το οποίο θα εκπροσωπήσει όποια πιο πολλές γίνεται. Το θέμα λοιπόν είναι πότε έχουμε ζημία σε περίπτωση στρέβλωση του ανταγωνισμού, στην αερομεταφορά, την ευρωπαϊκό συμφέρον και θα πρέπει να βρεθεί και μια ισορροπία για τις ε, διμερείς συμφωνίες που υπάρχουν και σε ό,τι αφορά ε, τους απαραίτητους μηχανισμούς παρέμβασης ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά θέματα, αλλά να αφήσω ίσως καλύτερα τους συναδέλφους από τις άλλες ομάδες να πάρουν το λόγο και να σας πω ότι αύριο θα έχουμε τη δεύτερη συνάντηση των σκιωδών και άρα είναι σωστή η χρονική συγκυρία για τη συζήτηση αυτή που θα κάνουμε σήμερα σε ό,τι αφορά και την εξεύρεση συμβιβασμών. Ευχαριστούμε τον κύριο Πίπερ και θα δώσω το λόγο στην κυρία σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ήταν αναμενόμενο, πολλοί συνάδελφοι έχουν υποβάλει τροπολογίες που δείχνει πόσο σημαντικός είναι αυτός ο κανονισμός. Βρίσκω θετικό ότι οι περισσότεροι θέλουν ε, ε, έναν αποτελεσματικό κανονισμό ε, που θα προστατεύει τον σχετικό τομέα. Δυστυχώς όμως ε, υπάρχουν ε, και ε, συνάδελφοι οι οποίοι θέλουν να αποδυναμώσουν τον κανονισμό αυτό, ιδιαίτερα όσον αφορά τον αθέμητο ανταγωνισμό. Σίγουρα υπάρχει σημαντικό περιθώριο για την εξέβρεση συμβασμών. Είναι βέβαιη ότι ο κύριος Πίπερ θα επιδιώξει να υπάρξουν τέτοιες συμβαστικές προτάσεις. Το θέμα όμως είναι ότι με κάποιες τροπολογίες η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή δεν θα έχει καμία δυνατότητα να ε, να ε, αντιμετωπίσει περιπτώσεις του ανταγωνισμού. Ελπίζουμε όμως κάτι τέτοιο να μην χρειαστεί και το κείμενο από μόνο του να αποτελέσει φόβητρο. Δεν θέλουμε πάρα πολύ μακριέ προθεσμίε. Ε, ούτε όμω να είναι ε, ε, υπερβολικά σύντομε, ώστε να μην μπορεί να υπάρξει μια σωστή διαδικασία. Επίσης σημαντικό είναι να μπορέσει να ολοκληρωθεί το παράγωγο δίκαιο και να μην μας εμποδίζουν οι διακοπές για παράδειγμα διότι και αυτό θα είναι προς όφελος όλων των συμμετεχόντων όσον αφορά τα πρότυπα τρίτων χωρών δεν θα πρέπει να ισχύσουν για τις τρίτες χώρες πρότυπα που δεν ισχύουν ήδη και για μας. Θέλουμε λοιπόν να διατηρήσουμε έναν υγιή ανταγωνισμό, θέλουμε να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή αεροπλοεία και δεν θα πρέπει να βλάψει ο κανονισμός αυτός τους κατασκευαστές αεροπλάνων αλλά ούτε και να είναι εις βάρος των επιβατών. δεν θα πρέπει να αφήσουμε να μας εκβιάσουν μεγάλα ή μικρά τρίτα κράτη. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να έχουμε κατάλληλα μέτρα προστασίας. Ευχαριστώ. Η κυρία Φώστερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Μόλις λάβαμε κάποιες συμβαστικές προτάσεις από τον κύριο Πίπερ, αλλά όπως υπόθηκε έχουμε συνάντηση των σκιωδών αύριο το πρωί έχουμε κάποιες σημαντικές ανησυχίε όσον αφορά την συνολική κατεύθυνση. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή. φαίνεται ότι οι συνάδελφοι θέλουν να καλύπτονται όχι μόνο οι αεροπορικές εταιρείες ε, αλλά ε, και οι ε, ρυθμιστές ενέργεια κυκλοφορία, ε, τα αεροδρόμια, οι κατασκευαστέ αεροπλάνων κλπ. Έχουμε όμω ε, νομοθεσία νομίζω που να καλύπτει όλους τους τομείς αυτούς. Εγώ είχα την εντύπωση ότι μόνο οι αερομεταφορεί μα ενδιαφέρουν εδώ και ότι υπάρχει άλλη νομοθεσία για του άλλου τομεί. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να έχουμε σχετική διευκρίνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή. Όσον αφορά την επίλυση διαφορών. Εγώ βλέπω να υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε διμερείς συμφωνίε και έναν κοινό ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Για παράδειγμα, αν υπάρχει διμερή συμφωνία ανάμεσα στη Γερμανία και κάποια χώρα του κόλπου, έχει ήδη συμφωνηθεί αυτό και υπάρχει ήδη εκεί μηχανισμό επίλυση διαφορών και αυτό θα είναι θέμα των δύο κρατών μελών. Και δεν βλέπω εδώ να έχει ρόλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι δεν πρόκειται για ε, συμφωνία Open Skies. Σε τέτοια περίπτωση ε, θα αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ο κύριος διαπραγματευτής εδώ. Τα κράτη-μέλη συμμετέχουν ε, ακόμα και όταν μιλάμε για το Open Skies, διότι ε, συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει διάκριση. Δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια διμερή συμφωνία. Δεν νομίζω ότι έχει αρμοδιότητα για κάτι τέτοιο και όσον αφορά τις επικρίσεις ε, που ακούστηκαν ε, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ε, θέσπιση κυρώσεων ε, ή ε, την απόσυρση θέσεων προσαπογείωσης, τα σλότς δηλαδή. Δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εδώ καμία αρμοδιότητα, διότι τα δικαιώματα αυτά είναι θέμα μεταξύ των κρατών μελών και όχι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν απονέμει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα σλότς. Θα ήθελα λοιπόν και εδώ διευκρίνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσπαθήσαμε να ε, φτιάξουμε έναν πιο σφιχτό κανονισμό αφαιρώντας διάφορες ε, τροπολογίες ε, και επίσης την δυνατότητα βλάβης διότι δεν θα πρέπει να μιλάμε για δυνατότητα, δεν πρέπει να μιλάμε για κάτι υποθετικό, θα πρέπει να έχουμε γεγονότα τα οποία να μπορούν να εξεταστούν. Και δεν εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή κανέναν άλλον ε, να ε, αρχίσει να προσπαθεί να αλλιεύσει στοιχεία λόγω Κάποιας, λόγω κάποιου ισχυρισμού. Άλλωστε έχουμε πολύ καλές εμπορικές σχέσεις με όλες τις χώρες με τις οποίες συνάπτουμε συμφωνίες. Και έτσι όπως διαμορφώνεται ο κανονισμός μπορεί τελικά να έχουμε μεγάλη ζημιά ε, πολύ εύκολα. Τελική παρατήρηση. Αύριο είπαμε θα έχουμε συνάντηση των σκιωδών. Ε, Ποιο είναι λοιπόν ο ρόλο του Κοινοβουλίου. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, μηχανισμό επίλυση διαφορών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάζει κάτι και να έχουμε πολιτική επιρροή. Δεν είναι δουλειά των Ευρωβουλευτών της Επιτροπής μας να έχουμε επιρροή σε μια υπόθεση ε, διμερή ανάμεσα σε δύο κράτη σχετικά με τα δικαιώματα. Θέλουμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ε, διευκρινίσει το θέμα αυτό. Θα πρέπει να επιβάλλει κυρώσεις. Αυτό νομίζω θα ήταν πολύ άστοχο. Υπάρχουν νομικοί περιορισμοί όσον αφορά ε, την ε, αποκάλυψη πληροφοριών από πλευρά ε, των επιχειρήσεων. Ούτε μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάει σε τρίτε χώρε και να απαιτήσει πληροφορίε σχετικά με τι επιχειρήσει τη. Μπορεί κάποιο να έχει την καλή βούληση να θέλει να μοιραστεί κάποιε πληροφορίε μαζί μα, αλλά δεν υπάρχει εδώ εξοεδαφικότητα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να περιορίσουμε το θέμα αυτό στην ουσία. Υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός στις ε, σχέσεις μας με άλλες χώρες. Ε, υπάρχουν συμμαχίες, μην το ξεχνάμε αυτό. Ή θέλουμε να απογειωθεί το θέμα αυτό σε μια στρατόσφαιρα που τελικά θα βλάψει το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δώσει την εντύπωση ότι δεν είμαστε ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις το, ε, ε, η πρόταση αυτή δεν καλύπτει μόνο τον αθεμητό ανταγωνισμό. Εγώ θέλω να έχουμε θεμητό ανταγωνισμό, απλά ανησυχώ διότι η έκθεση αυτή φαίνεται να παίρνει τελείω διαφορετική κατεύθυνση. Σα ευχαριστώ κύριε Στελίσκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Όπω είδαμε, Λάβαμε από τον κύριο Πίπερ τι πρώτες συμβαστικέ τροπολογίε. Ε, έγινε μια συζήτηση, θα γίνει μια συζήτηση αύριο και προφανώς θα πρέπει να καταβάλουμε μια προσπάθεια σοβαρή. Να περιοριστώ στι τροπολογίε και στη λογική κάποιων τροπολογιών. Η πρώτη παρατήρηση, αν θέλετε, Καταρχάς, νομίζω ότι πιστεύω ότι υπάρχει το θέμα της συμπληρωματικότητας των δύο εργαλείων της διμερής επαφές και την συμφωνία δηλαδή. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των αεροπορικών μεταφορέων. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, θα πρέπει να υπάρχει χρονοδιάγραμμα και αυτό μπορεί να κινηθεί παράλληλα με τις διμερείς ε, συμφωνίες, αλλά δεν μπορούμε να στέλνουμε το μήνυμα ότι ανεξάρτητα από το τι θα πετύχουμε στις διμερείς συμφωνίες, συνεχίσουμε. Μάλλον μπορεί να συνεχιστούν οι έρευνες για το αναρθωμένο 868. Αυτό θα πρέπει να είναι εκ παραλλήλου. Και αυτό για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στις διμερείς συμφωνίες, γιατί μπορεί κάποιος να πάει πιο αργά, κάποιο πιο γρήγορα και τελικά να, αποτελούν, να υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες. Δεν μπορούμε λοιπόν να αφήσουμε αυτό να βλάψει την Ένωση. Να υπάρχει συμπληρωματικότητα όμως και να τη σεβαστούμε. Κατά δεύτερον, ήθελα να το θέσω στο τέλος ε, το θέμα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Κάποιοι να θέλουν πιο υψηλό επίπεδο προστατευτισμού, κάποιοι άλλοι πιο χαμηλό. Αλλά αυτό στο οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουμε είναι το εξή. Οι διαδικασίες και οι διαπραγματεύσει θα πρέπει να γίνουν στο τεχνικό επίπεδο. Έχουμε ένα αρμόδιο όργανο και βασιζόμαστε στο εργαλείο εμπορική άμυνα. Το έχουμε ελέγξει σε θέματα Και θα πρέπει, πιστεύω, λίγο πολύ να ακολουθήσουμε τη φιλοσοφία αυτή, αλλά και τη διαδικασία. Ο τεχνικός χαρακτήρας, λοιπόν, πιστεύω είναι πολύ απαραίτητο. Ιδάλω, και το βλέπουμε, πιστεύω, εκτό του Κοινοβουλίου. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ στο ιστορικό του Κοινοβουλίου. Βλέπουμε ότι υπάρχει πολιτικοποίηση των ερευνών. Από τη μία λοιπόν ναι, σε ό,τι αφορά την έγκαιρη δράση, την προστασία, τη δέουσα επιμέλεια. Αλλά να ακολουθήσουμε και αυτό στο οποίο ειδικευόμαστε τώρα, σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα της Ένωσης. Το θέμα δεν είναι να ορίσουμε τα συμφέροντα της Ένωσης, είναι ορισμένα. Και πάλι Έχουμε σχετική νομοθεσία, αλλά θα πρέπει να δούμε τις διαδικασίες σε ad hoc βάση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καθορίσει το τι θα πρέπει να γίνει προκειμένου να ακολουθηθούν τα συμφέροντα της Ένωσης. Και για μένα το βασικό θέμα, πέρα από την ανταγωνισμό, το δίκαιο ανταγωνισμό, το άλλο θέμα το οποίο είναι σημαντικό. Συγγνώμη, έχασα τη σημειώση μου. Πέρα από τον ανταγωνισμό είναι το θέμα της συνδεσιμότητας. Γιατί αυτό που δεν θέλουμε να συμβεί είναι το εξής. Οι αερομεταφορείς να αρχίσουν να παίζουν οι μεγάλοι κατά των μικρών και των μεσαίων. Το βασικό λοιπόν θέμα είναι συνδεσιμότητα σε ένα δίκαιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτό λοιπόν να το έχουμε υπόψη μας. Κατά τα άλλα, ναι, υπάρχουν θέματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε, διαδικασία, χρονοδιάγραμμα και ούτω καθεξής. Αυτά είναι νομίζω εφικτά. Και νομίζω μπορούμε να λάβουμε και τα συμφέροντα του κλάδου και να πετύχουμε μια συμφωνία. Αλλά θα πρέπει να ακολουθήσουμε την φιλοσοφία, την ακαιρεότητα και το, αν θέλετε, παρελθόν του κοινωτικού κεκτημένου. Να μην ξεκινάμε να επαναφεύρουμε τον τροχό. Να έχουμε υπόψη επίσης τη συμπληρωματικότητα των δύο εργαλείων. Τα υπόλοιπα θα τα βγάλουμε πέρα. Και νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο το έργο μας ε, κοιτώντας και τις συμβαστικές τροπολογίες από ό,τι νομίζω ως τώρα. Ευχαριστώ. Σε αυτό το θέμα μας ενδιαφέρει να προωθήσουμε τον ανταγωνιστικότητα και τις, την ανταγωνιστικότητα και τους ίσους όρους ανταγωνισμού χωρίς να καταφύγουμε στον προστατευτισμό. Θα πρέπει να υπάρχουν ίσοι όροι για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, είτε είναι ε, ευρωπαϊκοί είτε όχι. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, συγκαλυμμένες επιδοτήσεις. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ε, δίκαιος και ελεύθερος ανταγωνισμός και θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής αυτού του ρυθμιστικού πλησίου. Ευχαριστούμε κύριε Νταλούντε. Και εγώ ζήτησα το λόγο. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει το λόγο, ας τον πάρω κι εγώ. Πριν δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Θα ήθελα να πω γενικά ότι πρόκειται για ένα μέσο άμυνας εμπορικού τύπου. Οι παρούσες διατάξεις ε, δεν είναι αποδοτικές και γι' αυτό χρειάζεται και αυτή η αναθεώρηση και γι' αυτό έχουμε και την έκθεση Πίπερ. Το μόνο πρόβλημα είναι, το μόνο πρόβλημα είναι μία ευαισθητοποίηση, γενικότερη ευαισθητοποίηση, αλλά πολλές φορές φτάνουμε σε κολυσιεργία και καταργούμε το ίδιο το διατακτικό του ρυθμιστικού πλαισίου. Για παράδειγμα, Επανερχόμαστε στις ε, διμερείς συμφωνίες, ε, αναστέλουμε ή παρατείνουμε τις προθεσμίες, όπως είπε και η κυρία Φώστερ. Υπάρχει ε, θέμα εξοεδαφικότητας. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει σωρία μέτρων και τρόπων όπου αναστέλλονται τα δικαιώματα του εμπορικού τομέα. Ε, χάρη όταν μιλάμε για ε, εξοεδαφικότητα στην Κίνα. Άρα απογυμνώνουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο. Το θέμα που τίθεται είναι της συνδεσιμότητας που ανέφερε ο συνάδελφος Βλέπουμε τι συμβαίνει. Τη στιγμή που δεν υπάρχουν ε, μεγάλοι κόμβοι στα αεροδρόμια, εκεί υπάρχουν ε, αντισταθμιστικά μέτρα ή αντίπινα μέτρα υποτύπων αντιπίνων κατά αυτών των εταιριών. Μας ενδιαφέρει λοιπόν η συνδεσιμότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προασπίζουμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα στον εμπορικό. Τώρα, ε, σε χώρες που δεν είναι διεθνής κόμβοι, θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα στο ιστορικό των κρατών μελών για τις δυνατότητες ε, συνδεσιμότητας παρά να θεωρήσουμε ότι τα συμφέροντα των ε, ε, εξωτερικών συνιστοσών επικρατούν επί των εσωτερικών. Γιατί η πρόταση γι' αυτό ακριβώς ε, προβάλλεται. Τη στιγμή που δεν υπάρχει συνδεσιμότητα, τότε καλύτερα να απομακρυνθούμε από αυτό το πλαίσιο. Ο κύριος Κορνέλης έχει το λόγο γιατί δεν τον ζητάει κανένα άλλος και μπορεί να λάβει το λόγο και η Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε και καλό σας απόγευμα. Πράγματι, αρκετές τροπολογίες έχουν υποβληθεί, τις εξετάσαμε με προσοχή. Υπάρχουν ορισμένες πολύ ενδιαφέρουσες για να ενισχύσουμε το κείμενο, διότι όπως είπε και, είπε και ο κύριος Ρικέ, μερικές κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση Γι' αυτό θα βρούμε έναν τρόπο ώστε να συμβαδίσουν αυτές ε, οι συνιστώσεις που κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση. Θα ήθελα να τονίσω τρία σημεία πέρα από τη συζήτηση που θα έχετε μεταξύ σας. Το πρώτο αφορά την, ε, τη λειτουργικότητα αυτού του μέσου θα πρέπει να ξέρουμε ότι ό,τι και να κάνουμε θα πρέπει να είναι λειτουργικό το πλαίσιο, αλλιώς δεν έχει νόημα. Και εδώ υπάρχει ένα σημείο που είναι νεότερο σε σχέση με τις προγενέστερες συζητήσεις που αφορά τις δραστηριότητες ή διαδρομές ή συμφορήσεις για τον ε, περιορισμό της εφαρμογής του κανονισμού, δηλαδή να μιλάμε αναζεύγει πόλεων. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι καλό, γιατί παραβλέπει την πραγματικότητα της ε, αεροπλοείας. Ξέρουμε ότι όταν πετάμε προς τις Ηνωμένε Πολιτείες δεν μιλάμε μόνο για άμεση μετάβαση Βρυξέλλες ΗΠΑ, μιλάμε για διάφορες διασυνδέσεις και γι' αυτό ε, αν μιλάμε για ζεύγη πόλεων τότε φτάνουμε σε μία ανελιξία η οποία δεν μας βοηθάει καθόλου. Πιστεύουμε ότι οι τροπολογίες 98 και 99 θα υποσκάψουν την χρήση του κανονισμού. Τώρα, ως προς τις διμερείς συμφωνίες των κρατών μελών, αυτό είναι πολύ σημαντικό στη συζήτηση, είχε συζητηθεί και στο Συμβούλιο Είχαμε ε, νομικές συμβουλές και από τη νομική υπηρεσία της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου που μας είπαν ότι ο κανονισμός είναι συμβατός με τις διμερείς συμφωνίες των κρατών μελών όπως έχουν επιτάπητος και επ' αυτού μας βοηθούν ορισμένες δικλίδες ασφαλείας. Δηλαδή κανένα μέτρο δεν μπορεί να ληφθεί που θα οδηγήσει στα κράτη-μέλη να παραβιάσουν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις και παράλληλα όταν ένα κράτος μέλος επιλύσει ένα θέμα δυνάμει της διμερούς συμφωνίας τότε η Επιτροπή θα πρέπει να το ελέγξει. Άρα αυτές οι δικλίδες ασφαλείας βοηθούν τα θέματα συμμόρφωσης μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και προστιθέμενη αξία γιατί πολλές διμερείς συμφωνίες ε, ε, σιγούν ως προς το θέμα της ε, ανοιχτής και ανταγωνιστικής αγοράς. Άρα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν ορισμένες πολιτικές και επίσης δεν υπάρχει θέμα επίλυσης διαφορών. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ κοντά ως Ευρωπαίοι έτσι ώστε να ε, προωθήσουμε και να λάβουμε υπόψη και τις διμερείς συμφωνίες, κάτι το οποίο γίνεται αποδεκτό από την ενιαία αγορά. Πιστεύουμε ότι η πρόταση της υποχρεωτικής ε, διεξοδικής χρήσης των μηχανισμών επίλυσης διαφορών πριν κάνουμε κάτι για αυτό τον κανονισμό, με αυτό τον κανονισμό δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Οι 28, 31, 58 και άλλες ε, τροπολογίες θα καταστήσουν αυτόν τον κανονισμό ε, καθόλου λειτουργικό και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για την ε, πραγματική χρήση των μέσων, όχι από πλευράς διεξοδικότητας. Τώρα, ως προς το θέμα της συνδεσιμότητας, και αυτό είναι ύψης της σημασίας, η συνδεσιμότητα για μας αποτελεί το επίκεντρο αυτής της πρότασης, θα πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε ανοιχτές και ανταγωνιστικές αγορές για να υπάρχουν πολλοί παίκτες και προσφορές. Πιστεύουμε όταν ε, εφαρμόζουμε αυτό το μέσον, όταν λαμβάνουμε μέτρα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή την ε, συνδεσιμότητα. Γιατί ε, αφορά τα κοινά συμφέροντα και φυσικά τα ευρύτερα οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Σε δύο φάσεις, πριν αρχίσουμε τις έρευνες και πριν λάβουμε μέτρα. Θα προβούμε στη δοκιμή, ε, δοκιμασία Ένωσης χωρίς να αποτελέσει ένα επιπρόσθετο κριτήριο για υποβολή καταγγελίας απλώς θα αφορά πρακτικές που προβαίνουν σε διακρίσεις και που στρεβλώνουν την αγορά. Αυτή θα πρέπει να είναι η βάση της καταγγελίας. Η συνδεσιμότητα δεν θα πρέπει να είναι, να είναι κριτήριο της καταγγελίας όπως ορίζει η τροπολογία 89. Τέλος, ως προς τη... τα θέματα χρονικών ορίων, θα πρέπει να έχουμε χρόνο για πραγματική έρευνα και να εξεύρουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ σπουδής, ποιότητας και ουσίες. Και τέλος, ως προς την τελική λήψη απόφασης, θεωρούμε ότι θα πρέπει να κρατήσουμε το ρόλο της Επιτροπής και έτσι θωρακίζουμε τα κράτη-μέλη κατά των πιέσεων από όπου και αν προέρχονται χρησιμοποιώντας τις αποφάσεις το, της Επιτροπής όπως χρησιμοποιούνται στο δίκαιο ανταγωνισμού. Και ελπίζω να γίνουν πολύ καλές συστήσεις αύριο μεταξύ ε, σκιωδών. Ευχαριστούμε κύριε Κορνέλης να δώσω πάλι το λόγο στον εισηγητή. Στον κύριο Πίπερ. Νομίζω ότι από την έκταση των σχολείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανησυχούμε. Κάτι χάνουμε μάλλον στο Κοινοβούλιο. Δεν πάση περιπτώσει, όχι καλά θα πάνε τα πράγματα. Να επισέλθω λίγο στα μεμονωμένα στοιχεία τα οποία έφτιαξαν οι συνάδελφοι. Συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Πρόης από τους Ασταλικές Δημοκράτες. Είπε ότι αποδυναμώνεται και ότι θα πρέπει να παραμείνει η αποτελεσματικότητα του, της ρύθμισης. Συμφωνώ με αυτά που είπε και το ECR ωστόσο, ότι δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε. Όπως είπε η κυρία Φώστερ, να δούμε ποιες είναι οι άμεσες δράσεις τις οποίες μπορούμε να δρομολογήσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε για να διαχωρίσουμε τα πράγματα και να μην υπησέλθουν τομείς της οικονομίας που δεν παίζουν κανένα ρόλο. Και σε ό,τι αφορά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ως Κοινοβούλιο Δεν συμφωνώ και εγώ να αναμειχθούμε στο πεδίο αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε λίγο πίσω και να δείξουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά θεωρώ ότι είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί, να έχει μάλλον τι απαραίτητε αρμοδιότητε, γιατί είναι καλύτερο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίζεται ω ένωση με κρατικές ε, οικονομίε. Ε, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είναι και αυταρχικές αυτές οι οικονομίες. Είναι καλό λοιπόν να βρούμε καλές λύσεις και όχι να κάθονται να ταλαιπωρούνται με μονομένα κράτη-μέλη από εταίρους που σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυσανάλογα δυνατοί. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να υπάρχει ευρωπαϊκό πλαίσιο. Να υποστηρίξω επίσης αυτά που είπε και ο συνάδελφος Τελίτσκα από την Άλντε. ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη υπερβολική πολιτική διάσταση. Να κοιτάξουμε το τεχνικό σκέλος και προς την κατεύθυνση αυτή να στείλουμε τέτοια μηνύματα. Κοιτώντας τα πράγματα με την ησυχία μας. Δεν χρειάζεται να τόσο μεγάλη αναστάτωση όσο είναι στην παρούσα φάση στα κράτη-μέλη. Επίσης, μου άρεσαν αυτά που είπαν και οι πράσινοι ίση όρια ανταγωνισμού. Αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να ακολουθήσουμε και αύριο στη συναντήση των σκιωδών και με βεβαίω ότι θα πετύχουμε καλούς συμβασμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πίπερ και να υπενθυμίσω ότι η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 20 Μαρτίου. Μάλιστα και συνεχίζουμε τις εργασίες μας, παραμένουμε στον τομέα των αερομεταφορών να ε, κάνουμε μια ανταλλαγή απόψη με την Επιτροπή σχετικά με την έκθεση για την ετήσια έκθεση του 2016 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 300 του 2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας. Ο κύριος Κάρλος Μες που είναι ήδη εδώ μην ακολουθήσετε το παράδειγμα του κύριου Κορνέλης. 5 έως 10 λεπτά σας δίνουμε. Και κύριε Κορνέλης, προφανώς και έβαμε. Ο κύριος Κάρλος, λοιπόν, έχει το λόγο. Εγώ τα άλλη φιλοδοξία δεν έχω σε αυτή τη ζωή, να κάνω να ακολουθήσω το παράδειγμα του κύριου Κορνέλης. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα σε όλους. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Νομίζω ότι το έγγραφο που έχετε μπροστά σας ε, είναι αυτονόητο. Ξεκινώντας από το άρθρο 16, ε, η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή υποβάλλει σε τακτικά, τα χρονικά διαστήματα έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του σχετικού κανονισμού και σας δίνει και μια εικόνα σχετικά με τις εξελίξεις στην ε, πολιτική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση για το 2016. Καταρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη διότι συνήθως η έκθεση αυτή υποβάλλεται νωρίτερα αλλά επειδή είχαμε εσωτερικό έλεγχο φέτος ε, αποφασίσαμε να περιμένουμε τα αποτελέσματα των εκθέσεων των κρατών μελών για να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε τα αποτελέσματα στο έγγραφο αυτό. Σίγουρα λοιπόν δίνει πιο σαφή η εικόνα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα δεδομένα που θα βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας 4 σχετικά με τα επίπεδα συμμόρφωσης. Σημαντικό είναι να επισημάνουμε ότι ένα από τα εργαλεία που έχει στη διάθεση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει ελλείψεις στο επίπεδο ασφάλειας είναι το άρθρο 15 που προβλέπει ε, να ε, βγει από τον ε, ε, από τον χώρο των ε, αεροδρομίων ε, με ενιαία διαδικασία. Πάντως δεν χρειάστηκε καμία κοινοποίηση του άρθρου 15. Όλες οι ελλείψεις καλύφθηκαν αμέσως, κάποιες που χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο καλύφθηκαν με κάποια μέτρα υποκατάστασης για κάποιο χρονικό διάστημα. Γενικά έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τα κράτη-μέλη και έχουμε αναγνωρίσει ε, την ε, αντιστοιχία, την ισοδυναμία των ε, προτύπων με κάποιες χώρες, για παράδειγμα οι Ηνωμένε Πολιτείες, Καναδά, Μαυροπούνια κλπ. Κάποια αεροδρόμια τα οποία ε, εντοπίστηκαν βρίσκονται στις Ηνωμένε Πολιτείε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι πολύ σημαντικός μας εταίρος. Φροντίζουμε να έχουμε συντονισμένη δράση απέναντι στη διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα όσον αφορά και τα μέτρα της ΙΚΑΟ. Το 2016 είχαμε υιοθέτηση του ψηφίσματος ε, του ε, ε, Συμβουλίου Ασφαλείας ε, του ΟΗΕ για την ε, ασφάλεια στις αερομεταφορές. Και είναι σημαντικό να το έχουμε αυτό κατά νου, διότι έτσι θέλουμε να διασφαλίσουμε την προσαρμογή των μέτρων, την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Καταβάλλονται και γενικότερα προσπάθειες εντός της ΙΚΑΟ με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις πολιτικές πρωτοβουλίες θα ήθελα να επισημάνω τις εργασίες που γίνονται στον τομέα των τεχνολογιών και τον οδικό χάρτη που διαμορφώνει τις εργασίες ε, στο πολύ σημαντικό αυτό θέμα, όπου έχουμε στενή συμμετοχή όχι μόνο των κρατών μελών, αλλά και ε, άλλων ε, εχόντων συμφέροντα. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να φροντίσουμε η τεχνολογία να παίζει το ρόλο που ζητάμε εμείς από αυτήν και όχι να ε, έχει τελικά ε, ε, δεσπόζοντα ρόλο. Τα θέματα στα οποία θα ήθελα να επικεντρωθώ είναι η προστασία των δημόσιων χώρων των αεροδρομίων λόγω και των επιθέσεων εδώ στις Βρυξέλλες πρόπες τον Μάρτιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό, διότι πώς προστατεύει κανείς έναν χώρο που πρέπει να είναι ανοιχτός, ελεύθερα προσβάσιμος. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιούνται διάφοροι τρόποι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ε, ανέλαβε δράση στο θέμα αυτό αναλύθηκε η κατάσταση και μάλιστα είχαμε και επικοινωνία με την Υπηρεσία Ασφάλειας ε, των Μεταφορών ε, των Ηνωμένων ε, Πολιτειών της TSA. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω εδώ. Σας παραπέμπω και πάλι στο έγγραφο το οποίο είναι αρκετά περιεκτικό και πολύ ευχαριστώ θα απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ο κύριος Μαρινέσκο έχει το λόγο. Thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχει μεγάλη σημασία αυτή η πτυχή της ασφάλειας και ο νέος βασικός κανονισμός ε, ασχολείται με αυτό. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις σε σχέση με την ε, δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού να ασχοληθεί με αυτή την πτυχή του ζητήματος. Θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή κατά πόσο γνωρίζει γιατί τα κράτη-μέλη αντιτίθενται στη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού σε αυτό το τομέα. Όχι όλους τις, τους τομείς ρύθμισης, αλλά τους περισσότερους. Γιατί ε, ε, μιλάμε για τρομοκρατικές επιθέσεις και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να έχουμε μια εναρμονισμένη προσέγγιση. Δεν λέω ότι θέλουμε κάποιος να είναι επικεφαλής ε, των ε, ελέγχων ασφαλείας να υπάρχει μια υπεραρχή, αλλά χρειαζόμαστε ανταλλαγές πληροφοριών για μέτρα τα οποία θα σχετίζονται με μια κοινή προσέγγιση. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε. Η κυρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Τα τελευταία χρόνια πράγματι έδειξαν ότι όσον αφορά την ασφάλεια των αερομεταφορών ε, σίγουρα πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Η πολιτική μου ομάδα και εγώ πρόσφατα επισκεφτήκαμε ε, το αεροδρόμιο των Βρυξελών ε, για να μας παρουσιάσουν αυτή τη νέα αντιμετώπιση της ασφάλειας. Αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στο θέμα της ποιότητας και της κατάρτισης του προσωπικού Γι' αυτό και μένα με ενδιαφέρει η εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά ε, το σύστημα Smart Security ε, φύση ασφάλεια στα αεροδρόμια. Από ό,τι κατάλαβα υπάρχει ανάγκη βελτιστοποίησης ε, των ελέγχων. Από την άλλη είναι κάπως προβληματικό να επιλέγονται οι επιβάτες που θα περνούν από επιπλέον ελέγχους. Ε, πόσο μάλλον ε, όταν λαμβάνατε υπόψη τους ε, και η συμπεριφορά τους στο διαδίκτυο για παράδειγμα ή οι αγορές που κάνουν. Στο τμήμα 1 μιλάτε για την αξιολόγηση αεροδρομίων τρίτων χωρών. Αναφέρεστε στο αεροδρόμιο της Τζακάρτα. Υπάρχουν σχετικά σχέδια για το εγγύς μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πλήση. Κυρία Φώστερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για την εισήγηση της ε, Ήμουνα. Ε, η αρχική εισηγήτρια μετά τις επιθέσεις της, 9, της 11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκτοτε είχαμε πολύ στενές επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά που κάναμε τότε νομίζω ότι πράγματι αποδείχτηκαν πολύ καλά Σημαντικό είναι όλες οι χώρες ε, της ΙΚΑΚ να ε, εφαρμόσουν τα σχετικά μέτρα και πολύ σωστά τώρα που είδαμε αλλαγή των απειλών είναι πολύ σωστό που επισημάνατε το θέμα αυτό της ασφάλειας των ε, περιοχών γύρω από το αεροδρόμιο. Το είδαμε τώρα και στη Ρωσία αυτό. θα πρέπει να γίνονται επιπλέον έλεγχοι στο προσωπικό και ε, το προσωπικό εδάφους ε, Είμαι βέβαιη ότι έχετε συζητήσει και εσείς το θέμα αυτό με τους Αμερικανούς ε, συχνά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ε, έχετε εργαστεί ε, επιμελώς. Από τη μία δεν θέλει κανείς να προειδοποιήσει ένα αεροδρόμιο σχετικά με έναν επικείμενο έλεγχο. Από την άλλη δεν θέλετε κιόλα να κλείσετε το αεροδρόμιο για να κάνετε τους ελέγχους. Και η τελευταία μου παρατήρηση έχει να κάνει με τον τρόπο αντιμετώπισης των επιβατών. Πράγματι, δεν προσπαθούμε να κάνουμε profiling των επιβατών. Είναι θέμα πολιτικής ορθότητας και Εγώ που προέρχομαι από τον αεροπορικό τομέα, ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό και απαιτεί και πάρα πολύ χρόνο. Με τους ρυθμούς που πηγαίνουμε θα μπορούσαμε να περνάμε από μαγνητική τομογραφία. Αυτός είναι πολύ καλός λόγος η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει και το σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, ε, μήπως θέλουν οι επιβάτες να υποβάλουν πρόσθετες πληροφορίες για να περνούν πιο γρήγορα από τους ελέγχους. Νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε δημιουργικά το πώς θα χειριστούμε το θέμα της ασφάλειας στα αεροδρόμια, διότι οι αερομεταφορές ε, τώρα πια έχουν γίνει μεγάλη ταλαιπωρία. Και ακόμα και για ανθρώπους που πηγαίνουν διακοπές, Ε, περνούν από τέτοια ταλαιπωρία. Και οι άνθρωποι ε, που έχουν καταστήματα στο αεροδρόμιο λένε χρειάζομαστε περισσότερου πελάτε και εγώ του λέω, αστειευόμενοι βέβαια, ότι δεν έχουν χρόνο γιατί περνάνε από του ελέγχου ασφαλεία. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε καλύτερου τρόπου, ε, θα πρέπει να βρούμε πιο προηγμένου τρόπου να το κάνουμε αυτό. Η τεχνολογία έχει να παίξει ρόλο, αλλά απαιτείται και πολιτική βούληση και ευφυα για να δούμε πώ θα προχωρήσουμε από εδώ και μπρο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με τον τρόπο που φτάσαμε μέχρι εδώ. Πάντως, ε, συγχαρητήρια Κομισιόν, κάνατε πολύ καλή δουλειά και με τις εθνικές αρχές ε, και έχετε όλοι μα την υποστήριξη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δεγκράντε έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, λυπάμαι που ε, ήρθα καθυστερημένα. Βρισκόμουν αλλού σε άλλη επιτροπή. Ε, ασχολούμαι για πολύ καιρό για αυτό το θέμα και ήμουν εισηγητής για τα σκάνερ όταν ε, αρχίσαμε να ασχολούμαστε με αυτό το ζήτημα. Ε, ε, δεν έχουμε ανταποκριθεί στις ανησυχίες των πολιτών. Βεβαίως ε, ζήσαμε πολλούς κλειδονισμούς και ε, πλήγησαν και οι πολίτες. Έχουμε 60, ε, ε, έχουμε 60 εκατομμύρια πρόσφυγες ανά τον κόσμο, ανακύπτουν και οι τρομοκράτες, υπάρχει παγκοσμιοποίηση, πλήττονται οι γείτονε χώρες και η κινητικότητα δίνει πολλές ευκαιρίες σε πολλούς, αλλά αποτελεί και πρόκληση και αυτό που μας απασχολεί είναι η ασφάλεια πρωτίστως. Οι πολίτες φοβούνται τον, την τρομοκρατία και τους σχετικούς κινδύνους, αλλά δεν θέλουν οι πολίτες να περιοριστούν τα δικαιώματά τους. Οι αερομεταφορές θα πρέπει να είναι ασφαλείς και να μην υπάρχει ε, φόβος. Και φυσικά οι αερομεταφορές είναι η κορονίδα του γενικού μας, γενικότερου μελήματος αντιμετώπισης της ε, τρομοκρατίας. Η πρόκληση, η γενική πρόκληση είναι αυτή. Πώς ε, να εγγυηθούμε την ε, ασφάλεια χωρίς να πλήξουμε την κινητικότητα στα αεροδρόμια και στα σύνορα. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και η Europol μας μιλούν για νέα ε, μέσα δράσης της τρομοκρατίας. Και έχουμε και την ε, νέα πρόταση αιτίας. Τα κράτη-μέλη έχουν τα δικά τους τα εθνικά συστήματα PNR. Οι ευρωπαϊκές ε, αερογραμμές μιλούν για χρήση των προσωπικών δεδομένων, για καταγραφή τους. Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να είναι εύλογα, όπως και η διαχείριση των συνόρων και της μετανάστευσης. Η ασφάλεια στον ε, κυβερνοχώρο σχετίζεται και ε, ε, με, την, με τον χώρο των αερομεταφορών ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας στις Αερομεταφορές το τόνισε σε αυτό. Οι αερομεταφορές έχουν άμεση σχέση με την κινητικότητα αλλά και με τον πολλαπλασιαστικό κίνδυνο της διασποράς της τρομοκρατίας. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες ε, ως προς την πιστοποίηση ελέγχων ασφαλείας το Συμβούλιο μπλόκαρε την προσπάθεια αυτή. Η, η Επιτροπή ε, έχει αρχίσει εσωτερικές διεργασίες και θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή πρέπει να αλλάξει η στάση. Ξέρω ότι υπάρχουν δυσκολίες, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτά τα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες. Φυσικά θα χρησιμοποιήσουμε και την τεχνολογία. γιατί μας λέγεται ότι εντάξει δεν μπορούν να ψωνίσουν στο duty free οι επιβάτες γιατί φοβούνται τους ε, ελέγχους ασφάλειας, δηλαδή χάνουν πολύ χρόνο εκεί. Αυτό που έχει σημασία είναι να αξιόπιστη η έλεγχη. Ε, δηλαδή, σε αυτή τη διχοτόμηση ελευθερία ή ασφάλεια θα πρέπει να προσπίσουμε, να σταθούμε υπέρ της ασφάλειας, χωρίς να καταστήλουμε την ελευθερία. Πώς μπορούμε επίσης να προβούμε σε ανταλλαγή πληροφοριών. Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της τρομοκρατίας είναι η πληροφορία. Και όσες φορές δεν αποσοβήσαμε τους κινδύνους, αυτό έγινε γιατί δεν είχαμε αρκετές πληροφορίες. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να ξέρουμε πού υπάρχουν ε, δυσλειτουργίες στο σύστημα πληροφόρησης και τα σύγχρονα σκάνερ είναι ένας, και από τους, ένας από τους τρόπους αντιμετώπισης της ε, τρομοκρατίας. Δεν μπορούμε να θυσιάσουμε αυτά τα δεδομένα. Χρειαζόμαστε το PNR για να υπάρχει ασφάλεια. Γι' αυτό η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα για να προασπίσει, να υπερασπιστεί την ασφάλεια των πολιτών. Ευχαριστούμε τον κύριο Ντεγκράντε. Ο κύριος Κούν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό το οποίο διαρκώς ε, μας απασχολεί επί σειρά ετών ε, και στην Επιτροπή Μεταφορών σε ό,τι αφορά την ασφάλεια όλων των επιβατών, ε, όχι μόνο των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των άλλων πολιτών, το πώς μπορούν να μεταβούν από τα ένα δρόμο σε άλλο με ασφάλεια. Έχουμε πολλές εναλλακτικέ λύσεις που έχουμε συζητήσει ε, απαγόρευση των υγρών, σκάνερ σώματος, ε, προσωπικός έλεγχος, σωματικός έλεγχος, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει μητρό στο οποίο καταχωρίζονται ουδέτερος έλεγχος των ατόμων. Ανεξάρτητος. Πολλά έχουμε πετύχει εντοπιστές ε, μετάλλου, εκρηκτικών ουσιών, μπορούμε και αυτά να τα εισαγάγουμε με τεχνικές ε, λεπτομέρειες και η σύσταση των υγρών στο μεταξύ μπορεί να ελέγχεται με πολύ ενδιαφέρουσες τεχνολογικές εξελίξεις αλλά αυτό που είναι απαραίτητο πιστεύω είναι να γίνονται και δειγματοληπτικοί έλεγχοι και να υπάρχει και ένα profiling όπως κάνουν και άλλες χώρες. Αυτό δεν πρέπει να το παραμελήσουμε κυρίως σε ό,τι αφορά τις ε, συνδυασμένες πτήσεις επιβάτες μαζί με εμπόρευμα. Και αυτό αποτελεί ξεχωριστό παράγοντα, τον οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και εδώ οι δύο αισθητήρε θεωρώ ότι παίζουν σημαντικό ρόλο. Το ξέρει και η κυρία Φώστερ, το K9. Έχει ως μονάδα εκπαιδευμένους σκύλους όπως το Gaulle για παράδειγμα, στο τμήμα των εμπορευμάτων, των εμπορευμεταφορών, όπου γίνεται δειγματοληπτική έλεγχη για... για μένα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε το εξή. Ότι υπάρχει και ο έλεγχος ε, ατόμων για τους προσωπικό, για το προσωπικό εδάφους. Και αυτοί είναι εξίσου σημαντικό να ελέγχονται για να μην αποτελούν ε, κίνδυνο. Άρα ναι, το προσωπικό αφενός και από την άλλη φυσικά και οι προμηθευτές. Οι προμηθευτές, ναι, αυτό έψαχνα. που δίνουν, για παράδειγμα, που φέρνουν ε, διάφορα αγαθά, duty free, δεν ξέρω και εγώ τι. Και εδώ θα πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρχουν ε, κενά στην ασφάλεια. Αυτά συνολικά. Νομίζω ότι προχωρήσαμε πολύ. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις, πολύ απλά ε, ε, εμφανίζονται ε, δίθεν τρομοκράτες με ένα πακέτο στην τσέπη τους. Και το προσωπικό θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο το τι να κάνει, το τι να κάνει. όχι μόνο δηλαδή στη εξαγωγή ελέγχων. Να υπάρχει, για παράδειγμα, ένας μικρός ε, γύρος, ένας μεγάλος γύρος ελέγχου γενικό και ένα μικρό για θέματα τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα. Ε, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκθεση. Έχει πολύ μεγάλη επιπτώσει γιατί θα πρέπει να ενισχυθεί και η εμπιστοσύνη των πολιτών. Να ξέρει ο πολίτης ότι όταν μπαίνει σε ένα αεροπλάνο είναι ασφαλή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κούν. Και για να δω ο κ. Κάρλος Μέστ αν θα ήθελε να απαντήσει και να εξαγαγεί συμπεράσματα για τα θέματα τα οποία ακούσαμε. 5-10 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Νομίζω ότι φτάνουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια από τα θέματα που αναφέρθηκαν, για παράδειγμα, σε σχέση με την ΕΑΣΑ. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι η ΕΑΣΑ έχει να παίξει ρόλο ιδιαίτερα όσον αφορά τον ε, σχεδιασμό της ασφάλειας ε, και πιστεύουμε ότι όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα κράτη-μέλη παίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Του του λεχθέντος δεν νομίζω ότι υπάρχει σημαντική αντίσταση, αλλά υπάρχει η αίσθηση ότι κάποια θέματα ασφάλειας από έκνομες ενέργειες ε, έχουν να κάνουν με πληροφορίες εμπιστευτικέ και ανήκουν μάλλον στον τομέα των ε, μυστικών ε, πληροφοριών. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με την ασφάλεια από φυσικές καταστροφές και όσον αφορά τον ε, βασικό κανονισμό, ήδη έχουμε ξεκινήσει διάλογο με την ΕΑΣΑ για να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα και να διασφαλίσουμε τα στοιχεία της ασφάλειας όπου η ΕΑΣΑ να μπορέσει να μας βοηθήσει να διοχετευτούν σωστά και να ε, εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες. Νομίζω λοιπόν ότι βελτιώνεται η κατάσταση. Επιτρέψτε μου επίσης να αναφερθώ στο θέμα των περιοχών γύρω από το αεροδρόμιο. Ε, ε, οι σχετικές επιθέσεις που είδαμε έχουν ε, προσελκύσει το ενδιαφέρον μας στο θέμα της ασφάλειας επιβατών και προσωπικού. Και δεν υπάρχει μία ενιαία λύση, δεν θα βρείτε εύκολα τεχνολογία που να μπορεί να βρει που να μπορεί να αποτελέσει ενιαία λύση. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια ε, πολυτομεακή προσέγγιση με διάφορα στοιχεία. Ένα από αυτά είναι η γενική νοοτροπία. Όχι μόνο το προσωπικό αλλά και το κοινό θα πρέπει να γνωρίσει το ρόλο που μπορεί να παίξει στην διασφάλιση της ασφάλειας. Επίσης ε, πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών όχι μόνο κατά τη διάρκεια και μετά από μία επίθεση αλλά και πριν. Ε, επίσης ε, θα πρέπει να είναι σαφείς οι διαδικασίες, να γνωρίζουμε ε, ποιος θα δίνει εντολές σε περίπτωση κάποιας επίθεσης. Επίσης θα πρέπει να προστατεύσουμε, θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στον αέρα. Στο Ζάβεντεμ ένα από τα πρέτα μέτρα που ελήφθησαν ήταν ε, να αυξήσουμε τη διάμετρο, να γίνουν ε, κάποιοι έλεγχοι λίγα μέτρα ε, έξω από το αεροδρόμιο. Αλλά αυτό δεν αποτέλεσε ικανοποιητική λύση. Θα πρέπει να έχουμε ροή επιβατών που να αποφεύγει που να αποτρέπει οποιαδήποτε συγκέντρωση επιβατών που μπορεί να γίνει στόχος τελικά. Επίσης, κυρία Φώστερ και κυρία Τεκράντες, Ε, το θέμα των εσωτερικών ε, απειλών. Η έλεγχη ε, του παρελθόντος των εργαζομένων, για παράδειγμα, είναι μόνο μία λύση και πάλι χρειαζόμαστε μία πολυτομεακή προσέγγιση. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μία ενιαία λύση. Θα μπορούσαμε όμως να βρούμε ένα σύστημα το οποίο να μας δώσει αυτά που θέλουμε και να φροντίσουμε να γίνεται αποτελεσματικός ε, έλεγχος των κινήτρων οποιοδήποτε εργάζεται στο αεροδρόμιο ή εργάζεται για κάποιον ε, ε, υπεργολάβο. Επίσης, στον κύριο Κούν να πω ότι σίγουρα το προσωπικό εδάφους περνάει από ελέγχους όπως και οι εταιρείες που εφοδιάζουν το αεροδρόμιο. Υπάρχουν λοιπόν σχετικά συστήματα, τα οποία όμως ενδεχομένως ε, να πρέπει να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε. Νομίζω ότι μια μάλλον φιλοσοφική συζήτηση που διεξάγεται αυτή τη στιγμή και απαντώ στην κυρία Φώστερ είναι το τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή δεν είναι βιώσιμη διότι θα δούμε αύξηση της κίνησης, αύξηση των επιβατών. Κάποιοι σαρωτές ε, μπορούν να αποτελέσουν λύση, αλλά οδηγούν και σε προβλήματα και ενδεχομένως και σε κάποιες αυξημένες τροτότητες. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να γίνει πολύ προσεκτικά και γι' αυτό ε, έχουμε ε, στενή συνεργασία με τα αεροδρόμια, με τις διάφορες ομάδες συμφερόντων, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα λειτουργικό. Το ίδιο ισχύει για την χρήση των πληροφοριών. Γνωρίζετε ότι οι κανονισμοί μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο αυστηροί από ό,τι σε άλλες περιοχές του κόσμου. Πρέπει να επαγρυπνούμε και να φροντίσουμε ε, να εκμεταλλευτούμε τις πληροφορίες αυτές ε, στον τομέα της ασφάλειας και να μην επιτρέψουμε σε ανθρώπους με κακούς σκοπούς να μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της κυβερνοασφάλειας. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και δεν αφορά μόνο τον ε, τομέα των μεταφορών, ούτε μόνο τον τομέα των αερομεταφορών. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε ό,τι έχουμε στα χέρια μας σήμερα. στο πλαίσιο της ε, οδηγίας, για παράδειγμα, και να δούμε τι συγκεκριμένες δράσεις θα μπορέσουν να ωφελήσουν τις αερομεταφορές και τι συγκεκριμένα μέτρα θα πρέπει να υιοθετήσουμε. Όσον αφορά την πιστοποίηση του εξοπλισμού ασφαλείας, ελπίζουμε να προχωρήσουμε γρήγορα και να βρεθεί η λύση που να μας επιτρέψει να προχωρήσουμε γρήγορα πάνω σε ένα θέμα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η ανταλλαγή πληροφοριών ε, είναι ένας τομέας που αναπτύσσεται πολύ θετικά και οι αξιολογήσεις κινδύνου αποτελούν τώρα πια ρουτίνα. με συμμετοχή των υπηρεσιών των κρατών μελών. Αυτό είναι ένα τομέα που θα συνεχίσουμε να εξερευνούμε και όπου θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μέστρα για αυτές τις διευκρινήσεις. Πρόκειται για την απαρχή αυτής της διαδικασίας και θα επανέλθουμε αγαπητοί συνάδελφοι λύεται η συνεδρίαση και θα τα πούμε τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου από τις 3. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα και ελπίζω να βρεθούμε σε κάποιο διάδρομο. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.